Let's begin, please. Buenos días. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε αυτή την έντονη ημέρα φορτισμένη με πολύ έργο. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ξέρετε ότι θα διεξαγάγουμε σήμερα το πρωί αυτή την ακρόαση για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα από τα στοιχεία της σημερίσιας διάταξης θα είναι η παρουσία του είπα του εκπροσώπου πριν, ε, των Ηνωμένων Εθνών, ο πρίγκιπας Σουσέιν, δεν μπόρεσε να προσθέτει διότι ακυρώθηκε η επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Θα προσπαθήσουμε να ξαναπρογραμματίσουμε αυτή την επίσκεψη μελλοντικά. Πρακτικά της 10 ε, ε, του, του Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αν δεν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, θεωρείται ότι κυρώνονται, την κρίνονται. Και ξεκινάμε έτσι τη συνεδρίασή μας. Συμφωνείτε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε συνέλθει εδώ για να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε κάπως τα πράγματα για ένα θέμα επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε κατά το παρελθόν ήδη και επί του οποίου πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις εργάζονται σε αυτό το θέμα. Και τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται και συνδέονται με το, τα Ολυμπιακά αθλήματα και τον αθλητισμό αφορά το θέμα αυτό τον σεβασμό των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Με συνοδεύει σήμερα το πρωί η συνάδελφος και φίλη Σίλβια Κώστα, πρόεδρος του, της Επιτροπής Πολιτισμού στο Ευρωκοινοβούλιο, που την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία της τη θετική της ε, προσέγγιση για να μπορέσουμε αυτό το έργο να το καλύψουμε από κοινού. Υπάρχουν και μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού που μας παρακολουθούν και είναι μαζί μας σήμερα. Το έργο συνεργασίας μεταξύ των διαφορών κοινοβουλευτικών επιτροπών θεωρώ ότι είναι θεμελιώδος σημασία. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου τη Επιτροπή Πολιτισμού το ότι για το ότι βρίσκονται εδώ σήμερα και για τη συνάδελφο Σίλβια Κώστα που επιθύμησε να προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία μαζί μα, Μια πρωτοβουλία που δεν θα παραμείνει μόνο στο πλαίσιο αυτό, στη δουλειά που θα κάνουμε σήμερα το πρωί, θα ακούσουμε πολλούς πραγματογνώμονες, ε, άτομα με μεγάλη ευαισθησία και γνώσεις γύρω από αυτό το θέμα. Θα τους ακούσουμε λοιπόν. Ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή δεν είναι παρά μόνο να συντονίσω αυτή τη συζήτηση να δώσω τα χαρακτηριστικά της. Έχει υποχρέωση πιστεύω η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ανθρώπου παγκόσμια και τόσο περισσότερο και στις περιπτώσεις των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων που βασίζονται στην παρουσία και έχουν την απήχηση των μέσων ενημέρωσης ευρωπαϊκών και παγκόσμιων και πολλών πόρων που αφιερώνονται οικονομικών κονδυλίων, ιδιωτικών και δημοσίων σε αυτά τα αθλήματα. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας δεοντολογικός κώδικας στεναρός και αποφασιστικός για τη συμπεριφορά και τη στάση των πόλεων, των κρατών που φιλοξενούν αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα ώστε να είναι σεβαστές οι προδιαγραφές για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προασπίζει πρώτα απ' όλα και κύρια και να δίνει το πρότυπο και το καλό παράδειγμα σε αυτή τη δέσμευση. Δεν θα αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή εγώ εδώ. Θα, το, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Δίνω τον λόγο στην κυρία Σίλβια Κώστα για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία αυτή μια πρωτοβουλία την οποία κάνουμε από κοινού με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι δύο μας επιτροπές πολιτισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρώ ότι μπορούν να έχουν πλέον ένα κοινό πεδίο εργασίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αξίες που εκπροσωπεί ο αθλητισμός μπορεί να προωθήσει και να μεταλαμπαδεύσει ο αθλητισμός και πειράζουν πάρα πολύ και τις διεθνείς μας σχέσεις. Να ευχαριστήσω λοιπόν πολλούς συναδέλφους Τρούπελ, Τροπιέσκι, Πέκοφ, από την Επιτροπή Πολιτισμού, καθώς επίσης και τον συνάδελφο Ζαγοράκη, ο οποίος είναι και πολύ σημαντικός αθλητής όπως γνωρίζετε. Θεωρώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε αυτή την καταπληκτική συμμετοχή από την Επιτροπή Πολιτισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας πενθυμίσω κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία νέα αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, αυτό το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε soft ήπια αρμοδιότητα, γιατί βέβαια θέλουμε να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητος, από την άλλη όμως είμαι πεπισμένη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να αναλάβουμε σημαντικότατη δράση και η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασχολείται προφανώς και με τους νέους και με τον αθλητισμό, έχει μια σημαντικότατη λοιπόν αρμοδιότητα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Να σας ότι στο 165 άρθρο της Συνθήκης Λισαβόνας λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει το ευρωπαϊκό προφίλ του αθλητισμού, των σπορ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αθλημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση που μπορεί να λάβει ο αθλητισμό, καθώ επίση και τη σημαντικότατη διάσταση εθελοντισμού που μπορεί να έχει ο αθλητισμό. Για τα ζητήματα λοιπόν αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αποφανθεί και μάλιστα είχαμε ήδη ένα ψήφισμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Θα αναφερθούμε βέβαια σήμερα περισσότερο στη διεθνή διάσταση του αθλητισμού, γιατί πρέπει και για αυτή τη διάσταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί. Θέλουμε να αναφερθούμε λοιπόν σε κάποιε σημαντικότητε αξίε. Στο αρχικό ψήφισμα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίσαμε κάποια ζητήματα τα οποία θα θεωρούμε ότι είναι βασικότατα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτον, να καταφέρουμε να γνωρίσουμε ότι ο αθλητισμό αποτελεί καταπληκτικό μέσο για την προώθηση τη ειρήνη και του διαπολιτισμικού διαλόγου και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο διάλογο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και διεθνικός Έπειτα προωθούμε ή πρέπει να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τις αξίες του αθλητισμού και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει και κατά τρόπο πιο απαιτητικό όσον αφορά δηλαδή την νομοθεσία την οποία μπορούμε να εγκρίνουμε. Θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο το fair play, την ακαιρεότητα των αθλητών, την αλληλεγγύη, καθώς επίσης και το στυλ ζωή, τον τρόπο ζωής που θέλουμε να προωθήσουμε μέσω του αθλητισμού. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει και σήμερα είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς γιατί η διαφθορά αποτελεί ουσιαστικά καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να αναφερθούμε στα στημένα παιχνίδια, καθώ επίση και στα τελευταία ψηφίσματα του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει και εμεί να καταφέρουμε να εγκρίνουμε τα ψηφίσματα αυτά του Συμβουλίου τη Ευρώπη στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε φαινόμενα όπω το ντόπινγκ και αυτό το έχουμε τονίσει στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ επίση και το ρόλο του αθλητισμού για τη διαπαιδαγώγηση των νέων και το ότι ο αθλητισμός μπορεί να οδηγήσει τελικά σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να καταφέρουμε δηλαδή να αποτρέψουμε διάφορες ασθένειες μέσω του αθλητισμού. Μπορεί ο αθλητισμός να προωθήσει περισσότερο τη δημοκρατία, να μειώσει τις σειράξεις και τις συγκρούσεις και θα πρέπει επίσης να αφαιρθούμε και στο ζήτημα της διακυβέρνησης του αθλητισμού, στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικότερος πλουραλισμός. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στην αρχή των μη διακρίσεων. Είχα πάει στο Ιράν πριν από λίγο καιρό και ουσιαστικά θα θέλαμε σε χώρες όπως το Ιράν ή για πράγμα στο Κατάρ αναφερόμαστε πολύ συχνά για το ποδόσφαιρο και τη διοργάνωση του ε, Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Θα θέλαμε λοιπόν, και αυτό είναι το όνειρό μας κατά κάποιο τρόπο, να μπορούν και άλλες χώρες όπως το Ιράν, το Κατάρ αλλά και χώρες της περιοχής αυτής να μπορούν περισσότερο να συμμετέχουν σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις έχοντας όμως παράλληλα μια πολύ σημαντική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν και οι νέοι από τις ε, χώρες αυτές και οι γυναίκες από τις χώρες αυτές να μπορούν να συμμετέχουν στα αθλήματα χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού που αναφέρεται στη συμμετοχή των νέων στα πλαίσια των αθλητικών διοργανώσεων και αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στο ζήτημα του αθλητισμού στα πλαίσια του προγράμματο Εράσμου. Το δικαίωμα λοιπόν στον αθλητισμό θα πρέπει να γίνει ένα δικαίωμα αναγνωρισμένο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και θα πρέπει όλοι να μπορούν χωρί διακρίσει να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Θέλουμε λοιπόν εμείς ε, σήμερα να αναφερθούμε στη διεθνή διάσταση του αθλητισμού και να καταφέρουμε να εντάξουμε τον αθλητισμό σε αυτό το οποίο ονομάζουμε πολιτισμική διπλωματία. Ο Μπάνκι Μουν πριν από λίγο είπε ότι ο αθλητισμός είναι μια γλώσσα που όλοι μας μιλάμε. Είναι ένα σημαντικότατο μήνυμα αυτό στα πλαίσια λοιπόν της πολιτισμικής διπλωματίας, την οποία θέλουμε εκ νέου να προωθήσουμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Θέλουμε ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η παιδεία αλλά και ο και ο αθλητισμός κυρίως διαδραματίζεται σημαντικότατο ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς μπορούμε μέσω του αθλητισμού να προωθήσουμε όλα τα δικαιώματα αυτά που άπτονται του αθλητισμού. Και σύμφωνα με τον Διεθνή Χάρτη για τον Αθλητισμό και την Παιδεία της UNESCO, ο αθλητισμός θα πρέπει να προωθήσει περισσότερο τη δημοκρατία καθώς επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη βία. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό το χάρτη που αναφέρεται στα δικαιώματα αυτά. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Μπακού που θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τους αγώνες αυτούς στα πλαίσια του Ολυμπιακού Χάρτη και του θεματολογίου του Ολυμπιακού 2020 να έχουμε συγκεκριμένε ρήτρε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την ευκαιρία των αγώνων αυτών ελπίζω ότι θα επιβεβαιωθεί πραγματικά έμπρακτα ο χάρτη αυτό και νομίζω ότι όλο και περισσότερο από κοινού θα πρέπει να ασκούμε πίεση προκειμένου ο οποιαδήποτε χώρα ή πόλη φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά γεγονότα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πολύ σημαντική ρήτρα για την επιλογή, ως πολύ σημαντική προϋπόθεση για την επιλογή συγκεκριμένης, συγκεκριμένης πόλης για τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Το Σεπτέμβριο επίση θα έχουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τον Αθλητισμό και ήδη από τώρα θα ήθελα να προτείνω δύο πράγματα. Η Επιτροπή Πολιτισμού θα διοργανώσει ένα workshop την επόμενη εβδομάδα από τι 7 έω τι 12 δηλαδή. Θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και θέλουμε να εορταστεί η εβδομάδα αυτή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια του workshop που θα διοργανώσουμε θα θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ε, παιδείας καθώς επίσης και της ε, σωστής εφαρμογής των αρχών που θα πρέπει να διέπουν από τον αθλητισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε επίσης και μια έκκληση προς ε, όλα τα κράτη-μέλη αλλά και προς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να έχουμε την κατάλληλη νομική βάση που ήδη υπάρχει προκειμένου να προσχωρήσουμε στη Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν έχουν υπογράψει ακόμα αυτή τη σύμβαση καθώς επίσης και το ψήφισμα 2014 του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει να κάνει με την ε, κατάχρηση, χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων. Αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι οι ομοσπονδίε ε, ποδοσφαίρου όπως η FIFA φέρουν προφανώς μια σημαντικότατη ευθύνη για την πρόθεση βέβαια του αθλήματος αυτού και είναι πολύ σημαντικό οι ομοσπονδίε αυτέ να προωθήσουν τι αρχέ τι οποίε πρεσβεύουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προσέγγιση λοιπόν αυτή, με την ολική, με τη σφαιρική αυτή προσέγγιση, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να προωθήσουμε τελικά την κατάλληλη πολιτική, την οποία ήδη έχουμε αρχίσει να προωθούμε εμεί στην Επιτροπή Πολιτισμού. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν στου προσκεκλημένους μα. Νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική εκπροσώπηση και του κόσμου του αθλητισμού και των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων των πιο σημαντικών. Ξεκινάμε δίνοντας τον λόγο στην κυρία Μίκη Βόρντεν, Διευθύντρια της Global Initiatives και Human Rights Watch. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ έρχομαι από τη Νέα Υόρκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλου ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί αυτή τη σημαντική συζήτηση σε μια κρίσιμη φάση για, παγκοσμίως για τον αθλητισμό. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν ήδη οι δύο συμπρόεδροι και θα σας πω ότι είμαι οπαδός του αθλητισμού. Μας αρέσει δε σε όλους να βλέπουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να βλέπουμε τους τελικούς, να υποστηρίζουμε τις ομάδες μας και χαιρόμαστε όταν οι σπουδαίοι μας αθλητές πάνε τα ρεκόρ. Όμως όλο και πιο δύσκολο γίνεται αυτό. Οι οπαδοί του αθλητισμού δεν θέλουν να κάθονται σε ένα στάδιο όπου χρησιμοποιούνται ε, και εργαζόμενοι που δουλεύουν υπό άθλιες συνθήκες. Εδώ ο δίπλα μου ο Φλόριαν Μπάουερ, ο αθλητικογράφος, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει ούτε παρενόχληση, ούτε λογοκρισία, ούτε να φοβάται να καλύψει κάποιο αθλητικό γεγονός. Οι δε ακτιβιστές οι οποίοι παρουσιάζουν τις καταχρήσεις γύρω από τον αθλητισμό θα πρέπει να τιμωρηθούν. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση. Οι διακρίσει είναι μια άλλη κατάχρηση που υποβαθμίζουν ε, το δίκαιο αγώνα, τους κανόνες του αθλητισμού και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές χώρες έχουν υποχθόνους νόμους που, που, που προωθούν τις διακρίσεις ή είναι εις βάρος των αθλητών LGBTI. Οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία δεν μπορούν να αθληθούν, ούτε γίνεται φυσική αγωγή στα κρατικά σχολεία και είναι αυτό θέμα εθνικής πολιτικής. Ο Ολυμπιακός Χάρτης όμως λέει πως ο αθλητισμός είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Όταν όμως δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να αθληθούν ή όταν συλλαμβάνονται επειδή προσπαθούν να παρακολουθήσουν κάποιο διεθνές ε, τουρνουά σε ένα στάδιο όπως στο Ιράν, θα πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν το κύρος μας, το κύρος μας ώστε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Η Human Rights Watch εδώ και πάνω από μια δεκαετία παρακολουθεί την, κατά, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και διαφόρων ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουμε εδώ μια σειρά από δημοσιεύσεις, όπως αυτές εδώ, που καλύπτουν αυτές τις παραβιάσεις ή καταχρήσεις από την Κίνα στη Ρωσία, από τη Σαββική Αραβία στο Κατάρ. Έχουμε καταγράψει πώς τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα επιφέρουν μεγάλες παραβιάσεις όταν ε, γίνονται, ανατίθεται η διοργάνωση των αγώνων σε ε, καταχραστές των ανθρωπίνων σαουδικη Γίνεται κατάχρηση μεταναστών, εργατών που χτίζουν τα στάδια, ε, ε, επιδεινώνεται το περιβάλλον, αποκλείεται η κοινωνία των πολιτών, υπάρχουν διακρίσεις και αποκλεισμοί. Καμία κυβέρνηση δεν είναι τέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμω η Human Rights Watch δείχνει από τι εκθέσει μα ότι οι καταχρήσει και οι παραβιάσει γίνονται ακόμα χειρότερε όταν οι διοργανωτέ είτε οι ίδιοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε το κράτο δεν είναι κράτο δικαίου εκεί που ανατίθεται η διοργάνωση. Και γιατί θέλουν όλα τα κράτη να διοργανώνουν ε, τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Γιατί, γιατί ε, φαίνεται η χώρα τους, ε, προκαλείται, προσελκύεται η προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα σπουδαία αυτά αθλητικά γεγονότα και όχι στο τι συμβαίνει στη χώρα. Κατασκευάζουν τεράστιες εγκαταστάσεις και αυτή η τάση αμφισβητεί την ηγεσία του αθλητισμού αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα έτος ε, φέτος όπου οι υποσχέσει αυτές θα δοκιμαστούν από κάποιου από τους χειρότερους παραβιαστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε κάποιες ημερομηνίε κλειδιά για να παρακαλώ βάλτε τα στα ημερολογιά σας. 29 Μαΐου η FIFA θα εκλέξει νέο πρόεδρο. Ο σημερινό πρόεδρο προσπαθεί για πέμπτη φορά να εκλεγεί, ενώ υπάρχουν προκλήσει ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια και το μεταρρύθμιση για τα εργατικά δικαιώματα. Όποιος αναλάβει τη FIFA θα πρέπει να ασχοληθεί με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάχρηση των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών, όπου, ε, όπως στη Ρωσία ή στο Κατάρ, όπου με το σύστημα γνωστό ως καφάλα ε, ε, γίνεται τρομερή κατάχρηση. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι είναι αποκλειστικά εργαζόμενοι εκεί. Τώρα, επίσης Αντί επίσης για τα, το, τα παιχνίδια της, ε, της ε, του Μπακού, υπάρχει και γίνεται ε, καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Ο πρόεδρος Αλία έχει συλλάβει δημοσιογράφους και, και ακτιβιστές οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να παρουσιάσουν το τι γίνεται. Τους έχει βάλει όλους φυλακή οι ηγέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μικρό κανάλι, ε, αυτό το μικρό παράθυρο πριν την έναρξη των παιχνιδιών για να επιμείνουν για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα αυτή. Οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές και η οργάνωση της Ρώμης που αποτελείται από 25 τέτοιες επιτροπές έχει την εξουσία να απαιτήσει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων ε, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν να ξεκινήσουν οι ε, αγώνες. 30 Ιουλίου τώρα. Καζακστάν και Κίνα θέλουν να φιλοξενήσουν τους ε, χειμερινούς αγώνες του 2030 και οι δύο χώρες είναι καταπιεστικές, αυταρχικές, πατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Καζακστάν δε έχει ένα, σύντομα μπορεί να έχει τον ίδιο νόμο με τη Ρωσία όσον αφορά τους ανθρώπους LGBT το να μάθουμε τα διδάγματα του Πεκίνου και του Σότσι σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται ε, στους όρους ε, στους όρους ε, σεβασμού των ανθρωπίνων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 15, ε, μάλλον 4 Αυγούστου θα έχουμε ένα χρόνο μέχρι Σότου να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο της Βραζιλίας. Ε, η Σαουδική Αραβία ακόμα δεν έχει επιτρέψει γυναίκες να συμμετέχουν, ε, ούτε καν στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα πρέπει να πάρουν το χρυσό μετάλλιο επειδή κατέφεραν να στείλουν μια αποκλειστικά αντρική ομάδα στους ασιατικούς αγώνες και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να... Και, και μάλλον και ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν έτοιμες οι γυναίκες αθλήτριες. Και φυσικά πώς να είναι έτοιμες αφού δεν επιτρέπουν στις γυναίκες τον αθλητισμό καθόλου. Κάθε μια από αυτές τις ημερομηνίε λοιπόν που σας ανέφερα ε, αποτελούν μια δοκιμασία για το παγκόσμιο αθλητισμό. Εμείς είμαστε μέλος ε, της ε, Διεθνούς Συμμαχίας για τον Αθλητισμό, μιας συμμαχίας ε, κοινωνία των πολιτών που θέλει να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, στη διάρκεια των μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Πιστεύουμε ότι όταν οι αθλητικοί οι διοργανωτές ε, σιωπούν ή όταν χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τις χώρες που διοργανώνουν τους αγώνες, αυτό υποβαθμίζει τους, ε, τα ίδια τα θεμέλια του αθλητισμού. Για πολλά χρόνια διεθνεί ε, αθλητικοί οργανισμοί όπω η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αθλητισμό. Και όντω δεν θα πρέπει να ασκούνται πιέσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα γύρω από τι αθλητικέ διοργανώσει. Όμω, όταν όλο ένα και περισσότερε καταπιεστικέ και αυθαρχικέ χώρε υπόσχονται ότι δήθεν θα σεβαστούν τον Ολυμπιακό Χάρτη, ε, ότι θα, θα, θα, ε, πραγματικά γίνεται η κατάσταση εφόρητη. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και ε, δεν χρησιμοποίησε πάντοτε αυτό το κύρος της. Οχτώ μήνες πριν από το Σότσι η Ρωσία υιοθέτησε τους, ε, τον νόμο περί των LGBT. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να πιέσει ώστε να απορριφθεί ε, χρησιμοποιώντας τον αρχή 6 του Ολυμπιακού Χάρτη για την μη διάκριση. Αλλά δεν έκαναν τίποτα τελικά. Με τα κοινωνικά μέσα η προσέγγιση της Διεθνούς ε, Ολυμπιακής Επιτροπής έχει αλλάξει και αν εφαρμοστεί θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για όλα τα σώμα, τους οργανισμούς διεθνού αθλητισμού. Ζήτησε, ζητήθηκε από τις ε, διάφορες ε, Ολυμπιακές πόλεις να σεβαστούν τον Ολυμπιακό χάρτη όπως την ισότητα των φύλων, την, την απουσία διακρίσεων, αρχή 6, καθώς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά ε, καθιερώνονται από τις, την Ολυμπιακή Συνθήκη. Μετά από την μεγάλη απογοήτευση του Σότσι, ο πρόεδρος Μπακ υποστήριξε ότι θα πρέπει κάθε συμφωνία για ανάθεση Ολυμπιακών Αγώνων να διέπεται από όρους για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την απογοήτευση των Ολυμπιακών του Σότσι. Και καθώς επίσης ότι οι, προηγου... οι προηγουμένως μυστικές συμβάσεις με τις πόλεις τώρα θα, ήταν, θα δημοσιοποιούνταν. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ε, τους όρους ε, όσον αφορά τη συμφωνία περί ε, διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και για όσους δεν τηρούν τους κανόνες η τιμωρία θα πρέπει να είναι να, μην, να, να, να απορρίπτονται από την Ολυμπιακή οικογένεια. Αν θες να συμμετέχει θα πρέπει να τηρήσεις και τους κανόνες. Ο πρόεδρος ε, ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια, αλλά με τις καταχρήσεις που γίνονται γύρω από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα πρέπει πλέον η Ολυμπιακή Επιτροπή να θίξει το θέμα αυτό γέρο πριν τον Μπακού και για τη FIFA να προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 12 δις κόστησαν οι Ολυμπιακοί του Πεκίνου και 57 οι Ολυμπιακοί του Σότσι. Και πολλοί πίστεψαν ότι αυτό ήταν ε, το περισσότερο που μπορούσε κανείς να δαπανίσει. Όμως ε, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί 2 εκατομμύρια από εκτιμούμε ε, ε, μετανάστες εργαζόμενους, θα, το κόστος εκεί θα ανέλθει στα 200 ε, εκατομμύρια δολάρια έχουμε υπολογίσει. Υπάρχει τεράστιο κόστος λοιπόν. Πολλοί ε, δε από αυτούς τους εργαζόμενους που εργάζονται υπό αυτό το σύστημα καφάλα όπως είναι γνωστό στο Κατάρ πέθαναν και χρειάζεται διαρκώς να έρχονται και άλλοι εργαζόμενοι από τον Νεπάλ και άλλες χώρες ε, της περιοχής. Μέχρι στιγμή οι ενέργειε που έχουν γίνει δεν αρκούν. Όσον αφορά το καφάλα, είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε καταναγκαστική εργασία. Το κατάρα απλά αλλάζει το όνομα, δεν κάνει καμιά σημαντική αλλαγή όμω στο ίδιο το σύστημα. Όσον αφορά τις θεωρήσει εξόδου, το κατά δεν έχει καταργήσει τον έλεγχο το εξόδου των εργαζομένων, ακόμα και όταν το αυθεντικό ε, προβαίνει σε καταχρήσεις. Η FIFA έχει ακόμα το χρόνο για να κάνει το σωστό, μπορεί και θα πρέπει να επιμείνει όσον αφορά την κατάργηση της άρνησης ε, θεωρήσεων εξόδου. Ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την σωστή μεταρρύθμιση, ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος καφάλα και μια διερεύνηση του γιατί πεθαίνουν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι, τόσοι πολλοί εργάτες. Κάποιοι θα σας πούνε ότι οι αθλητικοί οργανισμοί δεν έχουν κάνει μια εξουσία, και την πάση περιπτώσει δεν μπορούν να αλλάξουν ε, την εικόνα και το περιβάλλον. Αλλά αυτό δεν είναι νέο, αλλά ούτε και αληθινό. Μπορούν να ενεργήσουν ως μια πραγματική δύναμη ε, υπέρ του καλού. Στην ε, Νότια Αφρική, ας πούμε, δεν έχει γίνει ποτέ μια μεγάλη διοργάνωση λόγω του apartheid, λόγω του, των διακρίσεων η Ολυμπιακή Επιτροπή πίεσε την Βόρεια Κορέα να κάνει εκλογές πριν να αναλάβουν του, συγγνώμη, την Νότια Κορέα πριν να, αναλάβουν, να αναλάβει τους Ολυμπιακούς και έκτοτε είναι δημοκρατική αυτή η χώρα. Επίσης υιοθέτησε μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει το ντοπάρισμα, την περιβαλλοντικέ ε, τις επιρροές και αν δεν λάβουν κάποια μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταχρήσεις, θέλουν το, το λάθος μήνυμα στους καταχραστές, στους εκμεταλλευτές και θα ασκηθεί ακόμη περισσότερη πίεση σε αυτούς που ε, νομίμως ενεργούν. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση έτσι ώστε η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με την κρίσιμη στήριξη των Ευρωβουλευτών να χρησιμοποιήσετε το κύρος που έχετε ώστε να απελευθερωθούν στον Πακού οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές που είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Πλησιάζει η ημερομηνία γρήγορα. Δεν θα βοηθήσετε μόνο τους δημοσιογράφους του Αζερβαϊτζάν, αλλά και τους δικούς σας αθλητές. Κανένας δεν θέλει το μετάλλιό του να αμαυρωθεί από τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να πάψουν να ισχύουν διπλά μέτρα και σταθμά και να δίνονται οι διοργανώσεις μεγάλων αθλητικών γεγονότων σε διεφθαρμένες και αυταρχικές κυβερνήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να, πάψουν, να πάψει ο αθλητισμός να σχετίζεται με την κατάχρηση και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός μόνο για το καλό. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στη συνέχεια στον κύριο Μπάουερ που είναι δημοσιογράφος που έχει ειδικευτεί στα αθλήματα και στην πολιτική για τον αθλητισμό εντάξει την πολιτική για τον αθλητισμό. Για 12 λεπτά θα έχει τον λόγο. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τον χρόνο ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν οι ευρωβουλευτέ. Είναι λίγος ο χρόνος. Παρακαλώ να τηρήσετε τα όρια. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. <laughs> Δεν θα είναι πρόβλημα για μένα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν που με προσκαλέσατε. Θα ήθελα να σας εκπλήξω και να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι δεν θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα 12 λεπτά. Πρέπει τώρα να σας εκπλήξω γιατί έχασα τις σημειώσεις μου και δεν τις έχω εδώ. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να όσα θυμάμαι να σας τα αντλήσω από το νου μου και να σας τα παρουσιάσω και θα βασίζομαι στις ερωτήσεις και παρεμβάσεις σας υστερότερα. Αν παρακολουθήσατε τα επίκαιρα, είναι πολύ επίκαιρο αυτό το ζήτημα σήμερα και εγώ ίδιος ε, και όλες οι οργανώσεις μας ε, περνάμε μια ιδιαίτερα κέρια περίοδο και κατά τις πρόσφατες εβδομάδες όπου δημοσιεύθηκε χθες και προχθές δημοσιεύθηκαν αυτά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω οποιαδήποτε ερωτήματα θα είχατε στη συνέχεια. Τώρα, γενικά θα ήθελα να πω δεν θα υποβάλω κάποιες προτάσεις. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είναι δική μου δουλειά να υποβάλω προτάσεις. Μόνο κάποια σχόλια θέλω να κάνω για αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια τάση βλέπουμε, μια μετάθεση στα μεγάλα αθλήματα που πάνε σε αυταρχικές χώρες όλο και περισσότερο. Αυτό ξεκίνησε με τους Ολυμπιακούς του 2008 στο Πεκίνο και τις συζητήσεις που έγιναν γύρω από αυτό το γεγονός. Μετά είδαμε τα, α, τους Ολυμπιακούς στο Σότσι και μικρότερης εμβέλειας όπως για το χόκεϊ για παράδειγμα το διεθνές α, πρωτάθλημα στην Μπελαρούς ή κάποια χρόνια πριν όπως για το αφρικανικό κύπελο εθνών που έγινε στην Ισημερινή Γουινέα που έχει το μακρύτερο ιστορικό στην Αφρική όσον αφορά το αυταρχικό της ε, καθεστώς ε, και την καταπίεση, καταστολή. Και στο Σότσι οι αγώνες και όλες οι συζητήσεις που έγιναν δείχνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων που συνέβη εκεί, τα, τα προβλήματα που είχαμε όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, πολλές εφημερίδες ε, ε, και ε, άλλοι όπως και το International Human Rights και το Human Rights Watch ανέφεραν τα σχετικά και έγιναν και συζητήσεις για όλα τούτα. Και τελευταία, πριν από 4,5 χρόνια δηλαδή, από το κύπελο που δόθηκε στο Κατάρ, κύπελο ποδοσφαίρου, παγκόσμιο κύπελο, Όλα αυτά προκάλεσαν συζητήσεις. Ε, κοιτάζοντας γύρω μας ε, όσον αφορά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ποια είναι η απήχηση και τι συμβαίνει, υπάρχει και εκεί μια μετάθεση των πραγμάτων. Δεν έχουν επικεντρωθεί ουσιαστικά σε θέματα όπως τα, η την πολιτική και τον αθλητισμό ο αθλητισμός ήταν ένα θέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα που ήταν κάτι το οποίο αφορούσε την ευχαρίστηση των ε, ε, πολιτών, των ε, ανθρώπων και δεν θεωρείται ότι τα πολιτικά διαδραμάτισαν ένα μεγάλο ρόλο ούτε για τους ίδιους τους δημοσιογράφους ούτε για τον αθλητισμό. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε γενικά. Παρότι είδαμε μια μικρή μετάθεση, μια μικρή τάση στο διεθνή τύπο από τότε που αναφέρει αρκετές φορές τα θύματα που συζητούμε σήμερα, ο αγγλόφωνος τύπος για παράδειγμα, οι μεγάλες εφημερίδες όπως και το BBC εξάλλου και στη Γερμανία επίσης το έχουμε αυτό με ποιοτικέ εφημερίδες και τους δύο μεγάλους κρατικούς σταθμούς και το Deutschlandfunk ως εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό που αναλώνουν και επενδύουν χρήμα και χρόνο για να αναφέρουν αυτά τα γεγονότα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Επειδή είναι μέρος του γενικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Ότι τα μέσα δεν έδιναν μεγάλη προσοχή ή την προσοχή που θα έπρεπε σε αυτά τα θέματα ή αυτή που θα άξιζε την προσοχή, που θα άξιζε να τύχουν όλα αυτά. Στους διεθνείς οργανισμούς για παράδειγμα, που δεν θέτουν το πρόβλημα αυτό ε, σε σοβαρούς όρους και δεν το παίρνουν στα σοβαρά επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μετάθεση και τάση που είδαμε γιατί και πώς συνέβη στους διεθνείς οργανισμούς να δίνουν μεγάλα, μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις σε χώρες με αμφισβητήσιμο παρελθόν όσον αφορά την καταστολή και τον αυταρχισμό τους. Γιατί, πρώτον που θα έλεγα, πολλά πράγματα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν βέβαια. Μπορεί κανείς να ελέγξει και να αντιμετωπίσει κάποιους περιορισμούς ή να κάνει κανείς και του τους δικούς του νόμους. Αν δει κανείς για παράδειγμα τη FIFA 2018 ή προηγούμενα και κάποια νομοθετήματα τα οποία έγιναν και που παραβιάζουν θα έλεγα το διεθνές πλαίσιο της ε, νομολογίας ε, όσον αφορά αυτά τα θέματα. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτά τα αθλητικά γεγονότα για τις, τις διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς. Γιατί από πάνω προς τα κάτω είναι οργανωμένες και δομημένες αυτές οι οργανώσεις. Και ε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα σε λιγότερο δημοκρατικές χώρες ε, από πάνω προς τα κάτω. Επίσης, ε, όταν δει τις, τους Ολυμπιακούς που πρόκειται να διεξαχθούν και την απόφαση αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή όταν έρχεται η ώρα να βρει για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κάποιες χώρες που να είναι ικανές να συλλέξουν τα χρήματα, τα κονδυλία για να διοργανωθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Και τρίτον, ενώ αυτά τα θεσμικά όργανα τα οποία αναλαμβάνουν αυτά τα, αυτές τις εκδηλώσεις και τις δίνουν σε περισσότερο αυταρχικές χώρες, στο κάτω-κάτω είναι ο λογαριασμός. Πολλά περισσότερα χρήματα και κονδύλια ε, εμπλέκονται εδώ και πολλά, πολλά περισσότερα κέρδη μπορούν να, ε, να υπάρξουν. Και αν όλα αυτά τα συναθρήσει κανείς, όλα αυτά συναθρίζονται σε ένα ερώτημα. Δηλαδή, το θέμα της υπευθυνότητας, της ευθύνης. Αν δούμε λοιπόν ε, τις διάφορες πτυχές της ευθύνης και της υπευθυνότητας, βλέπουμε το διεθνές επίπεδο σαν, μια πρώτη, σαν ένα πρώτο πεδίο και προηγούμενα έχουν αναφερθεί θέματα σχετικά. Εγώ ίδιος το λέω αυτό το πράγμα και έχω αναφέρει τα σχετικά με γεγονότα τα οποία από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί. Αυτό το θέμα το αναφέρω και το θίγω σε κάθε δημοσίευμά μας όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί οι διεθνείς, διεθνείς οργανώσεις δεν υποχρεούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα θεωρούν ένα εκ προημίου ως προϋπόθεση ε, παράγοντα για διεθνείς τέτοιες ε, αθλητικές εκδηλώσεις. Κανείς ουσιαστικά και στο πολιτικό πεδίο δεν αμφισβητεί, δεν θέτει ερωτήματα και ζητήματα σε σχέση με αυτές τις ε, διεθνείς οργανώσεις. Και φυσικά υπάρχει εδώ εμπλοκή σε σχέση με τον αθλητισμό και, τον την πολιτική στα δύο επίπεδα. Αλλά τουλάχιστον ας πούμε το τι συμβαίνει και ας το δούμε. Για μένα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά σχεδόν δεν υφίσταται. Ενώ είναι η κατάσταση πολύ αμφισβητήσιμη. Δεν τίθεται ζήτημα. Και σε σχέση με τις μεγάλες τώρα οργανώσεις και η IWF, ε, όλες οι αθλητικές ε, ε, κοινότητες, καμιά από αυτές δεν έχουν θέσει προϋποθέσεις και όρους για τα δικαιώματα του ανθρώπου προκειμένου να κλείσουν κάποιοι αγώνες σε κάποια χώρα ως, ε, προϋπόθεση. Και αν δει κανείς τον κύριο Μπάχα, τον υπεύθυνο για τα όσα συνέβησαν για το 2020 στο Κατάρ, κοίταξα τα όσα αναφέρθηκαν, δεν βρήκα λέξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα άρθρο βρήκα, το νομίζω είναι στο 27 που τουλάχιστον αναφέρεται το θέμα της χρηστής διακυβέρνησης. Αυτό είναι όλο και όλο το οποίο αναφέρθηκε. Έχουμε αυτή τη μετάθεση πραγμάτων λοιπόν από τη μία πλευρά στην άλλη. Μία τάση λοιπόν όσον αφορά την προσέγγιση ε, σε σχέση με την διεθνή αθλητική ε, κοινότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν διαδραματίζουν ρόλο. Επειδή το κοινό όπως βλέπουμε κατά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αυτή την ε, ε, τάση που ακολουθείτε. Το κοινό δεν δέχεται πια αυτή την εξέλιξη και αυτή την τάξη πραγμάτων. Τι συμβαίνει με το Κατάρ για παράδειγμα. Ακόμα και προτού δοθεί στο Κατάρ. Και ποιος ε, είχε αναφέρει και ποιος είχε πει κατηγορώντας το Κατάρ ότι δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Αλλά επίσης αναφέροντας και για όλες τις προσπάθειες που είχαν γίνει. Το λέω αυτό επειδή ε, πρόκειται για κάποια χώρα που βλέπουμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, κοινή προσοχής εδώ και χρόνια. Και όλα αυτά τι μας δείχνουν. Μας δείχνουν σε σχέση και με τα όσα έγιναν στο Σότσι το πώς το κοινό, το κοινό και τα μέσα ε, παίρνουν αυτά τα μηνύματα και αντιδρούν και δρούν. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουν πολύ περισσότερο οι διεθνείς οργανώσεις αυτά τα πράγματα, ε, τα θέματα της χρηστής διακυβέρνησης και τα θέματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μειονοτήτων και ομάδων. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν τις χώρες ε, που ε, αναλαμβάνουν την εκδήλωση αυτών των αθλητικών γεγονότων. Εκτός από ίσως το Κατάρ, πέρα από αυτά δεν είδα πολλές εκδηλώσεις κατά τα τελευταία έτη όπου η δημόσια πίεση να έχει προκαλέσει κάποιες αλλαγές. Αυτές οι χώρες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχουν ευθύνες από πλευρά τους. Επίσης, είναι η ευθύνη να διασφαλίζεται η ελευθερία του τύπου, η, τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι σεβαστά, να μπορούν οι δημοσιογράφοι να επισκεφτούν αυτές τις χώρες και να δουν τι συμβαίνει εκεί, επιτόπου, να είναι σαφή όλα αυτά. Αν έχετε μια μεγάλη διάσκεψη, για παράδειγμα το Μάιο του 2014 στην Τόχα του Κατάρ, και όπου λέγεται ότι α, εντάξει θα αλλάξουν τα πλαίσια των δικαιωμάτων των εργαζομένων ε, ε αλλοδαπών εργαζομένων στο κατά... Ε, δίνεται συνέχεια μετά σε κάτι τέτοιο και αυτό κάναμε, δώσαμε συνέχεια, πήγαμε εκεί και είδαμε, ζητήσαμε να δούμε τι συμβαίνει και πολλοί δημοσιογράφοι από αγγλόφωνα μέσα και Γερμανοί, γερμανόφωνα μέσα δημοσιογράφοι ε, προσπάθησαν να, να διακριβώσουν τι γίνεται και επί τόπου και ακριβώς αναφέρθηκε, μας υποσχεθήκατε κάτι πριν από ένα χρόνο και τώρα τι θα κάνουμε. Ζητήσαμε κάποιες συνεντεύξεις εδώ και εβδομάδες πριν, εβδομάδε και εβδομάδε, Ζητήσαμε να μπορέσουμε να ε, δράσουμε και να πάρουμε εικόνες και να ε, ε, αναλύσουμε το τι γίνεται. Τι υπολογίζετε ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε επειδή δεν απαντάτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα και δεν μας δίνετε καμιά ευκαιρία. Θα το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε και εμείς ευθύνες και αυτό οδηγεί στο να αναλαμβάνουν τα μέσα τις ευθύνες τους και να είναι υπεύθυνα. Υπάρχει επίσης ευθύνη και υπευθυνότητα των μέσων και του τύπου και των δημοσιογράφων. Προέρχομαι από ένα τηλεοπτικό κανάλι που έχει κάποια κονδύλια για να επενδύει σε αυτού του είδους ε, τις εκδηλώσεις και πολλά, α, πολλοί άλλοι έχουν δυσκολίες. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετάθεση πραγμάτων, μια αλλαγή στην οτροπία δημοσιογράφων που θεωρούν τον εαυτό τους αθλητικούς δημοσιογράφους εντός εισαγωγικών ή μάλλον οπαδούς αθλημάτων και όχι πολιτικούς, πολιτικής ε, ε, ε, δράσεις ε, ή πολιτικής αντιμετώπισης δημοσιογράφοι που αντιμετωπίζουν τα αθλήματα υπό ένα πολιτικό πρίσμα. Λοιπόν, υπάρχει όμως ευθύνη και υπευθυνότητα από πλευρά των δημοσιογράφων να αναφέρονται αυτά τα θέματα, να καλύπτονται αυτά στις χώρες ε, περί των οποίων πρόκειται και να υπάρχει ευκαιρία που θα μας δίνεται για να καλύπτουμε αυτά τα γεγονότα όπως πρέπει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάου. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Φανή Μιχαλίδη που είναι υπεύθυνη για τα δημόσια θέματα της ε, Διεθνούς ε, Οργάνωσης Ποδοσφαίρου FIFA. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε της ε, Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, κυρία Πρόεδρε της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, την πρόσκληση αυτή την οποία απευθύνατε προς την FIFA και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε στη συζήτηση αυτή που διεξάγεται και να μπορέσουμε και εμείς να εκθέσουμε τις απόψεις μας όσον αφορά το σημαντικότατο αυτό ζήτημα, αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορούμε ως διοργανωτές σημαντικών αθλητικών γεγονότων να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο ιδίω τη διαδικασία επιλογή χώρα ή πόλη για τη διοργάνωση των αθλητικών αυτών γεγονότων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα να μπορούμε να συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση. Ανάλογη συμμετοχή είχαμε και στο παρελθόν όταν είχαμε πει ότι θέλουμε να συνεργαστούμε περισσότερο με τις κυβερνήσεις, με πολιτικές δημόσιες αρχές, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με επιστημονικά ερευνητικά κέντρα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να έχουμε και τη δική τους τη συμβολή. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι τομεί στους οποίους θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο, τις οποίες θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, ιδίω όσον αφορά τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ήδη και κάποια θετικά επιτεύγματα τα οποία συνδέονται με τον αθλητισμό και με τα αθλητικά γεγονότα και θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια τη συζήτηση και αυτά τα θετικά διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει. Κάλυψαν πολλά ζητήματα οι προλαλήσαντε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ήδη να δώσουμε κάποιε απαντήσει σε κάποια ερωτήματα τα οποία θέσανε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Ξέρω ότι μα πιέζει και ο χρόνο, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε και λίγο περισσότερο σε κάποια ζητήματα κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων που θα ακολουθήσουν των παρουσιάσεων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην αρχή να δούμε τι γίνεται με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και πώς διοργανώνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαιρικών Σωματείων, από την FIFA. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια σφαιρική παρουσίαση της διοργάνωσης αυτής, πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εφιστάμενα έγγραφα υποβολής υποψηφιωτήτων, γιατί ήδη έχουν ανεληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες για το ζήτημα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθώ και στη στρατηγική βιωσιμότητα που έχουμε. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ως οργάνωση για τη στρατηγική μας αυτή και θα ήθελα στη συνέχεια να κάνω και ένα σύντομο απολογισμό τις εργασίες που έχουμε επιτελέσει αλλά και τη πολιτική μα εργασία όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίω στα πλαίσια του παγκόσμιου Πρωτάθληματο ποδοσφαίρου τη FIFA όσον αφορά τη διαδικασία επιλογή πόλων και χωρών για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η FIFA τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ουσιαστικά μετα... μετασχηματίστηκε πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά αρχίσαμε να κάνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τη διακυβέρνησή μας. Είπατε κι εσείς ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Όντως αληθεύει αυτό και αυτός ήταν ο απότερος στόχος ο δικός μας. Αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε μέσω κάποιων τροποποιήσεων, αλλαγών, τις οποίες προτείναμε και εφαρμόσαμε σε διάφορους τομείς. Όσον αφορά την ηθική και τη διοντολογία που ακολουθούμε, όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής διαφόρων αποφάσεών μας, όσον αφορά την αλλαγή του καταστατικού μας, όσον αφορά την ε, διαδικασία εφαρμογής συγκεκριμένων αποφάσεων, την ε, αναθεώρηση των κανονισμών και των κανόνων, που έχουν να κάνουν με την διαδικασία την οποία ακολουθούμε για τον καθορισμό της πόλης ή της χώρας που θα αναλάβει την διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο επίπεδο εποπτείας παρακολούθησης και ένα καλύτερο επίπεδο λογοδοσίας. Γι' αυτό τον λόγο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε και την όλη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματο ποδοσφαίρου. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο ανοιχτέ διαδικασίε, έχουμε αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν και στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι αδυναμίες του παρελθόντος θα βελτιωθούν στο μέλλον ή θα ληφθούν τουλάχιστον υπόψη στις μελλοντικέ διοργανώσεις παγκοσμίων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέραμε όσον αφορά τη δικασία επιλογής είναι οι αλλαγέ που κάναμε όσον αφορά το σώμα εκείνο, το φορέα εκείνο που αποφασίζει για τη χώρα ή την πόλη την ευθύνη αυτή τη στιγμή φέρει περισσότερο το Κογκρέσο, αυτή η εκτελεστική επιτροπή της FIFA, η οποία θα ακολουθεί μια διαδικασία ανοιχτής ψηφοφορίας, ενώ την τελική απόφαση για, την, ε, για το διορισμό της πώληση της χώρας και αυτό θα γίνεται εντελώς ανοιχτά σύμφωνα με το άρθρο 80 του καταστατικού της FIFA όπου αναφέρουμε και τις ε, γενικότερες ε, παραμέτρους για την όλη διαδικασία διορισμού της ε, πόλης ή της χώρας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Όσον αφορά τώρα πιο ειδικότερα το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αυτό εστιαζόμαστε σήμερα στα πλαίσια της συζήτησής μας. Η δική μας η προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο στον βλέπουμε ως αποκλειστικό κριτήριο πώς έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια συγκεκριμένη χώρα. Στο μέλλον λοιπόν, οι επιδόσεις μιας χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να αποτελούν απαραίτητα φραγμό στην όλη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητος. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε γενικότερη τροχοπέδη στη διαδικασία επιλογής μιας χώρας και ουσιαστικά θα είχε αντίθετα αποτελέσματα από αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Θα ήταν ίσως και αντιπαραγωγικό. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια προσέγγιση κατάλληλη, ισορροπημένη, να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχουν οι, αθλητικές, ε, οι αθλητικοί φορείς. Αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στο ανθρωπιστικό δίκαιο και σαφώς θέλουμε να είμαστε και φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές, πραγματιστές ως προς το τι μπορούμε τελικά πραγματικά να πετύχουμε. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που έχουμε ως διοργανωτές αθλητικών γεγονότων για να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι χώρες που επιλέγουμε όντως τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η FIFA επί του παρόντος έχει ένα συγκεκριμένο δόγμα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιεί για την υποβολή υποψηφιωτήτων. Δεν έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά ε, τις μελέτες αντικτύπου τις οποίες διεξάγουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να βαθύνουμε περισσότερο σε αυτό το ζήτημα στο μέλλον. Ακόμα όμως και για τα έγγραφα υποβολής υποψηφιωτήτων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2022 υπήρχαν κάποιες πτυχές που είχαν να κάνουν με την ανθρώπινη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και προβλέπαμε συγκεκριμένε ρήτρε για τον ρατσισμό, την καταπολέμηση διακρίσεων και το καθεξής. Είχαν συμπεριληφθεί δηλαδή οι πτυχές αυτές σε διάφορα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιεί η FIFA, ιδίω στα πλαίσια τη διαδικασία υποβολή υποψηφιωτήτων. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλαμε να τονίσουμε ότι όντω μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ακαιρεότητα, η δεντολογική συμπεριφορά, η ε, βιώσιμη ανάπτυξη, η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε σχέση με όλα αυτά, θα πρέπει να αναφέρω και τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα. Για τη βιωσιμότητα με Θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ζήτημα αυτό γιατί είπαμε ότι ε, για κάθε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που θέλουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική βιωσιμότητα, ε, ακολουθούμε συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη, την ε, βιώσιμη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Ξέρετε ότι όλα τα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι δημοσιοποιημένα, είναι κείμενα στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Ξέρετε ότι τη στρατηγική αυτή ακολουθήσαμε και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Βραζιλία. Και νομίζω ότι στα πλαίσια των εγγράφων αυτών μπορείτε να δείτε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ακόμα και αριθμητικά δεδομένα, για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη η στρατηγική βιωσιμότητα της FIFA και τα επιτεύγματα στα οποία έχει οδηγήσει. Τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον όπως είπαμε και πριν από λίγο. Προσβλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ε, κατάρτιση των ε, απαιτήσεων για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιωτήτων για το 2022. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα πλαίσια του 2015, προκειμένου να επιλέξουμε την επόμενη χώρα που θα διοργανώσει τα αθλητικά γεγονότα του 2017 και θέλουμε να καταφέρουμε να δούμε ποια θα είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένε προϋποθέσεις που θα χρησιμοποιήσουμε. Ήδη το 2011 ο πρόεδρος της FIFA και ο γενικός γραμματέας της FIFA είχαν πει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους δύο αυτούς τομείς, βιωσιμότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά την διαδικασία επιλογής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και νομίζω ότι η δέσμευση αυτή που αναλάβαμε το 2011 αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή πολύ στεναρά στα όσα προτείνουμε. Δηλαδή, προτείνουμε μια προσέγγιση κατάλληλη, σωστή, ορθή, ισορροπημένη, που θα λαμβάνει υπόψη της διάφορες κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς που έχουμε λάβει από διεθνείς εξειδικευμένους φορείς στον τομέα του αθλητισμού και λαμβάνουμε προφανώ υπόψη μα και τόσα μα λένε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών. Και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη μα και τι νουθεσίε τόσο των κυβερνήσεων όσο και των δημοσίων αρχών. Σίγουρα το ζήτημα είναι αρκετά πολύπλοκο. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολε λύσει όσον αφορά τη διοργάνωση των μεγάλων αυτών αθλητικών γεγονότων, αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα δείτε κι εσείς όταν ξεκινήσει επισήμως η διαδικασία αυτή υποβολής υποψηφιωτήτων, όταν δημοσιοποιηθούν όλα αυτά τα επίσημα έγγραφα, θα εκπλαγείτε θετικά θεωρώ από τη νέα προσέγγιση την οποία ακολουθεί η FIFA και θα δείτε πόσο θαραλέοι και στεναροί είμαστε σε συγκεκριμένους τομείς. Το ότι θέλουμε πλέον να βελτιώσουμε πολύ περισσότερο την δέουσα επιμελητία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάλληλη διαχείριση, κατάλληλη αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ. Θα δώσω το πρώτο λόγο στο Μάρκ Τάιζεν. Δεν ξέρω αν πρόφερα καλά το όνομά σας. Τάιζεν, Τάιζεν, διορθώστε με παρακαλώ που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και την Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω ένθερμα ε, για την πρόσκληση που λάβαμε, δηλαδή όχι μόνο να συμμετέχουμε παθητικά σε αυτή την ε, ακρόαση γιατί πρόκειται για μια εκδήλωση όχι μόνο από αθλητικής άποψης αλλά και από πολιτικής άποψης πολύ σημαντική ε, και επειδή μπορούμε να εκφράσουμε τη σημασία που αποδίδουμε σε μια τέτοια συνεδρίαση αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αντιπροσωπώ ότι αντιπροσωπευόμαστε από τον αντιπρόεδρό μας Ζώνα Σκοτσιτσάνιτς αλλά και το Γενικό Γραμματέα του ΕΣΠΕ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής του Μισελ Φασπέρα που στη συνέχεια θα μπορέσει και ο ίδιος να απαντήσει σε ερωτήσεις γιατί σε αυτή τη μορφή μοιράσαμε κάπως την εργασία μας, την κατανομή εργασίας έτσι την κάναμε και είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας απευθύνω σήμερα το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου παρέμβαση με βάση κάποιες αρχές που είναι σημαντικό να πιστεύω να τις θυμίσουμε ώστε να μπορέσουμε να δούμε, γιατί άκουσα με πολύ προσοχή και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων σε αυτό εδώ το ε, στρογγυλό τραπέζι. Ε, ε, νομίζω πως είναι γενικός γεγονός και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ενώ πριν από κάποια χρόνια η πολιτική δεν υπήρχε, τα αθλητικά γεγονότα δηλαδή ήταν τελείως απολιτικά, ενώ πλέον και ο ίδιος ο πρόεδρος της ε, Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είπε ότι ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για να αγνοούμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά δεν είναι μόνο εκείνος που το είπε και ο προηγούμενος πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ιδιαίτερα στη διοργάνωση της, ε, των Ολυμπιακών του Πεκίνου, ε, έλεγε ότι ε, ακούμε διαρκώς το σφιγμό του κόσμου. Και Επίσης κάτι ακόμα που θεωρώ που είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ θύμισε και παραθέτω τα λόγια που είχε χρησιμοποιήσει ότι οι, τα ιδιωτικά των Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα ίδια με το ΟΗΕ, δηλαδή ε, η, ανοχή, η ισότητα και οι δίκαιοι αγώνες. Δυστυχώς όμως δεν το έχουμε καταφέρει πάντοτε. Ο πόλεμος ε, και η ε, δυσανεξία, η, ε, ξένους και εξακολουθούν να, επικρατούν στον κόσμο δυστυχώς ε, και γι' αυτό και ο αθλητισμός θα πρέπει να συνδεθεί με την πολιτική. Οι αθλητικές οργανώσεις ε, και οι διοργανωτές αυτών έχουν αυτό απολύτω συνειδητοποιήσει εδώ και κάποια χρόνια. Λαμβάνουν υπόψη τον τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό αντίκτυπο που έχει ο αθλητισμός, την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός στην κοινωνία μας, γιατί υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν έχουμε συζητήσει. Μιλήσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλήσαμε πολύ για διακρίσεις, αλλά πιστεύω πως ε, το κεφάλαιο το βασικό είναι η ε, κοινωνική ένταξη. Αυτό το διαπιστώνουμε στις κοινωνίες μας ε, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε πολλές χώρες όπου βλέπουμε το φαινόμενο της γλώσσας, το φαινόμενο των χρωμάτων, το φαινόμενο των διαφόρων πολιτισμών. Πιστεύω λοιπόν ότι ο αθλητισμός είναι ένα όχημα πολύ σημαντικό για την κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση και εκεί βεβαίως επηρεάζει και πολύ ε, τα όσα συζητήσαμε πριν από λίγο, δηλαδή τις διακρίσεις ή την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ε, δεν είμαστε εδώ βέβαια για να μιλήσουμε για άλλες πτυχές, ε, υγεία, πολιτική, παιδεία, αλλά περισσότερο για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε σχέση με τον αθλητισμό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεπερνούν ε, ε, τις διοργανώσεις ε, αθλητικών ε, γεγονότων. Πιστεύω λοιπόν πως σήμερα έχουμε προσκληθεί ως ένας θεσμός. Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή βρίσκεται εδώ για να συζητήσει μαζί τους και μαζί σας και είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας, όχι μόνο για να συζητήσουμε αλλά και για να αμφισβητηθούμε οι ίδιοι. Πρόκειται για μια πολύ θετική προσέγγιση που έχουμε λοιπόν απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και από την άλλη πλευρά και τα ακούσαμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αθλητισμός ως βήμα πολιτικής, αλλά θα πρέπει ωστόσο να βλέπουμε τι κάνουμε, από πού προερχόμαστε, από πού ξεκινάμε και δεν μπορεί να απαιτείται από μας να έχουμε εξουσία λες και είμαστε κυβέρνηση ας πούμε. Υπάρχουν οι κυβερνήσεις και είναι άλλος ο ρόλος τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμίσουμε. Ποια είναι η προσέγγιση που θα πρέπει να έχει ο αθλητισμός, δηλαδή μια προσέγγιση ουδέτερη που φυσικά δεν σημαίνει ότι ε, είναι α-πολιτική. Τώρα, μίλησα για κάποιες γενικέ αρχές Είπαμε ότι ωραία είναι τα λόγια και να, καλό είναι να είμαστε ανοιχτοί σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά συγκεκριμένα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε και πού οδεύουμε. Κάποια διδάγματα πρέπει να τα κρατήσουμε. Και όπως είπα, παρέθεσα και τον Τόμας Σεπά, θα πρέπει να δούμε τι έχει μεταφραστεί μέσα στην Ατζέντα 2020 και μια σημαντική συνέπεια είναι ε, το άρθρο 6 του Ολυμπιακού Χάρτη όσον αφορά την ανάθεση μεγάλων ε, αθλητικών ε, διοργανώσεων και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων δίνονται, ανατίθεται η διοργάνωση στις κάποιες πόλεις και από τη δική μας πλευρά θα πρέπει πάντοτε να σεβεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Βόρντεν για να παραθέσω ένα μόνο παράδειγμα μίλησε ας πούμε για τις διακρίσεις στις οποίες υπόκειται οι γυναίκες στην ε, Σαουδική Αραβία και στο Ιράν το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αλλά από την άλλη πλευρά ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και στο δικό μας επίπεδο το να παρέμβουμε ε, μπορούμε πολύ περιορισμένα ωστόσο στο παρελθόν υπήρξαν κάποια ανοίγματα και θα ήθελα να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Ζακ Ρόγκ ε, είχε προβεί σε τέτοιες συζητήσει με τον ε, πρόεδρο της Σαουδικής Αραβίας και ζήτησε και κατάφερε η μία γυναικεία ομάδα να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς στο Λονδίνο. Είναι ένα, μια μικρή, ένα μικρό στοιχείο, αλλά έγινε όμως. Πιστεύω πως όντως ένας από τους τρόπους για να παρέμβουμε δραστηρία είναι ε, η ανάθεση και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι πόλεις, Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, ε, ότι πρέπει να σεβαστούμε επίπεδα μισθών, συνθήκες εργασίας, θα πρέπει να διαπιστώσουμε την κατάσταση, ε, έχουμε την, το προνόμιο ε, και υπάρχουν διατάξεις στην Ευρώπη ε, όσον αφορά το εργατικό δίκαιο που είναι δημόσιες αυτές οι νομοθεσίες. Σε άλλες χώρες, δυστυχώς στις περισσότερες υπόλοιπες χώρες στον κόσμο δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα οι θεσμοί μας κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτό το πλαίσιο. Πρόσφατα ε, διάβασα ε, όταν υπήρχε μια ακρόαση, ε, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας είχε προσκληθεί, αλλά και αυτός διαπιστώνει ότι πρόκειται, εφόσον πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό που έχει κύρος και έχει δυνατότητες και εκείνο όμως περιορίζεται στις δυνατότητες παρέμβασης. Δεν μπορούμε να ζητάμε υπερβολικά πολύ κίνηση όσον αφορά τις ε, αθλητικές διοργανώσεις, αλλά στο επίπεδο του, της αρχικής συγγραφής υποχρεώσεων κατά την ανάθεση των αγώνων, ε, ε, θα, εκεί κάπως μπορούμε να επηρεάσουμε. Εξάλλου, ε, κάνουμε μια ολόκληρη σειρά συστάσεων ε, στις ε, πόλεις που είναι υποψήφιες για ανάληψη διοργάνωσης το των Ολυμπιακών, ας πούμε σεβασμός των, των αρχών του Ολυμπισμού. Απαγορεύονται οι διακρίσεις, όπως είπαμε, στο άρθρο 6, ε, επί τη βάση σεξουαλικών προτιμήσεων. Είναι κάτι το οποίο είπαμε με τη Σαουδική Αραβία, με τον προηγούμενο πρόεδρο της, Ευρωπαϊκ... της ε, ε, Ολυμπιακής Επιτροπής της Σαουδικής Αραβίας. Το γνώριζαν πάρα πολύ καλά, όμως υπάρχει και η κοινωνία γύρω από τη διοργάνωση. Δεν είναι πάντοτε εύκολο λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Κλείνοντας, επειδή τελειώνει και ο χρόνο μας, θα πρέπει να δούμε τις αθλητικές διοργανώσεις ως ένα όχημα το οποίο μεταφέρει τις κοινωνικές αξίες ε, ε, του δικού μας πολιτισμού. Επίσης και στο επίπεδο εκπαίδευσης, παιδείας είναι ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο. Στοιχείο πολύ σημαντικό όχι μόνο για, για τους νέους, και είμαι πεπισμένος ότι ο αθλητισμός είναι ένας από τους ε, ε, μία από τις συνιστώσεις στο πλαίσιο διαφόρων ε, φορέων και είμαστε φορείς κοινωνικών αλλαγών, είμαστε φορείς κινητικότητας ε, για τις κοινωνίες ε, και θέλουμε πάντοτε να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έλλειψη ή την κατάργηση των διακρίσεων. Αυτά είχα να πω στη συζήτηση τούτη. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Σάρα Βιτμάιερ που είναι επιστημονική συντονίστρια ενός προγράμματος ε, έρευνας του Ινστιτούτου Εξωτερικών μας Σχέσεων. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Βαλενσιάνο, αξιότιμη κυρία Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ο αθλητισμός μιλάει όλες τις γλώσσες, ε, συγκινεί τον κόσμο παγκόσμια ε, συνενώνει τον κόσμο και τους χαρίζει την ικανοποίηση κοινωνικά, γλωσσικά, πάνω από κοινωνικά, γλωσσικά ή πολιτιστικά εμπόδια. Στον σημερινό κατακαιρματισμένο κόσμο ο αθλητισμός μπορεί να είναι μια κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική δύναμη και έτσι να είναι ένα σημαντικό μέσο πολιτισμικών επαφών στην πολιτιστική διπλωματία στο πεδίο πολιτισ... του πολιτισμού για την ανάπτυξη και την εξασφάλιση της ειρήνης. Σε αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή στο έργο του More Europe Initiative και σε σχέση και με την ακρόαση, σε σχέση με τις Επιτροπές Πολιτισμού και Εξωτερικών το Μάτιο εφέτος. Το IFA, Ίδρυμα για τις Εξωτερικές Σχέσεις, είναι ένα μέρος του δικτύου για περισσότερη Ευρώπη. Το πρόγραμμα έρευνας εξετάζει επίκαιρα θέματα θέματα της πολιτισμικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε το δυναμικό για τις προκλήσεις για τον αθλητισμό στην εξωτερική ε, πολιτική και με την διάσκεψη πολιτισμός της δικαιοσύνης το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες με επιστήμονες και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σύντομα θα αναφερθώ στο δυναμικό του αθλητισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Η Μόνικα Σταμπ, πρώην προπονήτρια της ε, ομάδας γυναικών ε, του Κατάρ και ε, πρέσβυρα της Γερμανίας το 2014, ακολουθεί τέτοια προγράμματα ποδοσφαίρου με κορίτσια και γυναίκες σε πολλές χώρες του κόσμου, στο Πακιστάν, Ερυθρέα, Μπαχρέιν κτλ. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά ένα γήπεδο και μια μπάλα. Με πολύ λίγα κονδύλια μπορεί πολύ μεγάλη, ε, πολύ μεγάλη επίπτωση να επιτευχθεί. Έχουμε ίδια ευθύνη, έχουμε τα προγράμματα για το ποδόσφαιρο των γυναικών που μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα των γυναικών και να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να κατακτήσουν τις ελευθερίες τους. Η ενίσχυση του ποδοσφαίρου γυναικών θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των γυναικών στην κοινωνία. Όχι μόνο όσον αφορά την προαγωγή των γυναικών γυναικών αλλά και για τους ανθρώπους με μειονεξίες και ειδικέ ανάγκες και για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχολείο, στη γειτονιά, στην κοινωνία. Μπορεί ο αθλητισμός να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προαγωγή αξιών που θα εξυπηρετούν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ένα από τα μεγαλύτερα δυναμικά του αθλητισμού είναι η εμβέλεια που έχει φτάνει σε όλους τους ανθρώπους ε, όλων των ηλικιών. Με αυτό το εύρος ε, μπορεί ε, κοινωνίες και περιοχές που αντιμετωπίζουν σειράξεις και αναπτυσσόμενες χώρες να βοηθηθούν στην πρόοδό τους. Διευκολύνει έτσι τις επαφές ο αθλητισμός ποδόσφαιρο ή καποέρα στις τα προσφυγικά στρατόπεδα στο Λίβανο μπορούν να εμπλέξουν παιδιά και νέους ώστε να υπάρξει συζήτηση για την αποφυγή βίας και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Το δυναμικό του αθλητισμού στην αντιμετώπιση σειράξεων και τριβών στην κοινωνία πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική με την οικουμενικότητα των κανόνων, τις δοκιμασίες που συνεπάγεται για τους αθλούμενους και η σπουδαιότητα που έχει να είναι κανείς όπως του αθλητισμού δημιουργεί αξίες. Δημιουργούνται αξίες όπως ανεκτικότητα, αμοιβαία κατανόηση, συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών, πολιτικών συστημάτων. Στην εξωτερική πολιτική χρησιμοποιούνται τα αθλήματα ως μορφή για να προαχθούν όλα αυτά. Υπάρχουν και βιτρίνες χωρών μέσα από αυτές τις ε, δραστηριότητες. Μεγάλες λοιπόν εκδηλώσεις ε, μπορούν να ενισχύσουν ε, την εικόνα μιας χώρας. Συνεπάγονται όμως εδώ και κάποιες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2006 στη Γερμανία παγκόσμια βελτίωσε την εικόνα της Γερμανίας. Για την Βραζιλία για παράδειγμα έχουμε μια άλλη πτυχή όπου παρουσιάζονται πολλές φορές κοινωνικές ε, τριβές. Ε, αυτό το πρωτάθλημα, αυτά τα πρωταθλήματα κινητοποιούν χιλιάδες, μυριάδες πολιτών. Πολλές φορές ε, πρέπει να, τα προβλήματα αυτά να τα συνειδητοποιήσει κανείς. Έχουμε εδώ μια μεγάλη κοινή γνώμη που ασκεί κριτική πολλές φορές. Τα θλήματα αυτών των διαστάσεων είναι παιδεία, είναι σκηνές όπου μπορούν πολλά να προσφερθούν. Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες δράσεις προς τα έσω όπως για παράδειγμα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Σότσι. Τα όσα είναι, ε, είναι, έχουν αρνητική χρειά πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να συνειδητοποιήσει ε, το διεθνές κοινό αυτά τα προβλήματα. Κοινωνικές ανισότητες, παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου πρέπει να βρεθούν έτσι, βρίσκονται στο επίκεντρο. Με τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις ε, οι κοινωνικές και πολιτικές βάσεις πρέπει να συνειδητοποιηθούν και να διαδραματίσουν ένα ρόλο παγκόσμιες τέτοιες εκδηλώσεις είναι συναντήσεις κρατών, στρατηγιών, διεθνών οργανισμών, μια εμπλοκή πολλών εμπλεκόμενων από τα μέσα. Με την ανάληψη τέτοιων εκδηλώσεων πολλές φορές υπάρχουν και δεσμεύσεις χωρών όπως για παράδειγμα φιλελευθεροποίηση των αγορών. Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις που να μπορούν να συνδυαστούν με τέτοιες εκδηλώσεις. Μπορεί για παράδειγμα η ατζέντα, το θεματολόγιο 2020 του IOC να θεωρηθεί ότι πάει αρκετά μακριά. Διεθνείς τέτοιες οργανώσεις, διεθνείς ε, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνε για τη χρηστή διακυβέρνηση. Πρέπει οι στόχοι για την παγκόσμια ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών να ακολουθηθούν και να τηρηθούν ο Τζόζεφ Μαγκουάιερ, επαΐων της IFA και, του, και προγράμματος έρευνας στο Lockbury University του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να στοχεύουν σε ηθικούς προσανατολισμούς και κατευθύνσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θεσμικό όργανο ε, σφαιρικό που πρέπει να βασίζεται σε αξίες και αρχές που να διέπουν την εξωτερική της πολιτική, σεβασμός δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι εξαρτάται από αυτά τα στοιχεία η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ε, μεγάλης απήχησης παγκόσμια παρουσιάζουν και προβλήματα των κοινωνιών που αναδύονται στην επιφάνεια. Η πίεση είναι τέτοια ε, τόσο έντονη που πρέπει να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης των πληθυσμών επιτόπου. Για παράδειγμα στη Βραζιλία, αν υπήρξε μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων, μια απήχηση θετική δεν έχει ακόμα υπαρκώς αναλυθεί. Καταρχήν ωστόσο διαπιστώθηκε ότι μεγάλες τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις μόνο μια προσωρινή επιρροή έχουν στην ανάπτυξη μιας χώρας η δημοσίευση του οικονομολόγου Άντριου Τζίμπαλιστ με τον, με τον τίτλο Circus Maximus που το Φεβρουάριο του 2015 δημοσιεύθηκε <clears throat> δεν έχει κάποια οικονομικά κέρδη ε, που να διαπιστώνει για τις ε, επιμέρους χώρες μετά από τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις στην ε, Ινδία με, τα, με το Commonwealth Games του 2010 και την οικονομική ανάπτυξη για την απήχηση της Ινδίας Πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές ε, για την ε, συνέχιση αυτών των ε, εκδηλώσεων ώστε να υπάρξουν αηφόρες δομές στις χώρες αυτές προς την υλοποίηση αυτών των στόχων. Η τήρηση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η λογοδοσία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν συνάπτουμε συμβόλαια για την ανάληψη τέτοιων αθλητικών εκδηλώσεων από κάποιες χώρες. Οι ευρωπαϊκές αρχές αξίες πρέπει προς τα έξω να αντανακλώνται και πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνοψίζω, θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ότι η τεράστια εμβέλεια του αθλητισμού όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική κυβερνήσεων μπορεί να χαρακτηρίζει έθνη και κράτη, αλλά και γιατί ως μέσο της εξωτερικής πολιτικής έχει σπουδαιότητα ο αθλητισμός. Δημιουργούνται έτσι επαφές μεταξύ νεότερων και πιο ηλικιωμένων πολιτών, όλων των διαστρωματώσεων της κοινωνίας. διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να προαχθούν. Η δημοκρατία, η, το nation building, η δημιουργία, η ανοικοδόμηση κρατών, η η ολοκλήρωση, η κοινωνική ένταξη μπορούν να προαθούν. Ο αθλητισμός από πλευρά δυναμικού του πρέπει να ενταχθεί στην πολιτισμική πολιτική της Ευρώπης. Ενώνει τους πολίτες, δημιουργεί γέφυρες μεταξύ χωρών, δημιουργεί μια οικουμενική προσέγγιση και ενισχύει την εμπιστοσύνη. Θέλω να τελειώσω με αυτό που είπε ω παράθεμα Όρχαν Παμούκ. Το ποδόσφαιρο είναι πιο γρήγορο από τι λέξει από τα λόγια. Ευχαριστώ. Bueno, ah, muy bueno. Ahora voy a dar la palabra a nuestro colega Tarabella, que es el copresidente. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάρκ Ταραμπέλα, συνάδελφο, που είναι α, πρόεδρος της ομάδας Intergroup για τον αθλητισμό και μετά θα συνεχίσουμε δίνοντας το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν. Συνάδελφε Ταραμπέλα. Καλημέρα σας, ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι όντω συμπρόεδρος του Intergroup για τον αθλητισμό. Ο άλλος πρόεδρος είναι ο κύριος Φίσας. Αναγνωρίστηκε η νέα αυτή διακομματική ομάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι Καταρχάς να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Πολιτισμού αλλά και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διοργάνωσε αυτή τη σημαντικότητα δημόσια κρόαση για τον αθλητισμό, μεγάλα αθλητικά γεγονότα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ και εγώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλέκεται περισσότερο σε ζητήματα αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον έχει έναν επίτροπο ο οποίος ασχολείται ξεκάθαρα με ζητήματα αθλητισμού. Με τον Σαντιάγκο Φίσας εξ αρχής θελήσαμε να δημιουργήσουμε την διακομματική αυτή ομάδα, το Intergroup, στην αρχή τη νέας κοινοβουλευτική θητείας. Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θεωρήσαμε λοιπόν για αυτό το λόγο ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς ο αθλητισμός. Η διακομματική αυτή ομάδα, το Intergroup αυτό, ασχολείται με διάφορες πτυχές του αθλητισμού. 70 περίπου είναι οι ευρωβουλευτέ που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή. Συμμετέχουν και γυναίκες, όχι πάρα πολλές, αλλά η συμμετοχή τους είναι σημαντική και απαρτίζεται επίσης από πρώην αθλητές ιδιαίτερα ψηλού επίπεδου, ο Θοδωρής Ζαγοράκης ο οποίος είναι παρόν, πρώην επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας που κέρδισε το πρωτάθλημα το Ευρωπαϊκό του 2004 και ο κύριο Βέντα, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές του handball και με την Τζούντι Γκέρλινγκ, τη Βυζινή Ροζιέρα το Σαντιάνκο Φίσα και τον υποφαινόμενο αποτελούν το Προεδρείο αυτό του Intergroup. Από τα θέματα που θέλουμε να προσεγγίσουμε είναι ο αθλητισμός και η υγεία. Το να καταφέρνουμε να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, η σωματική άσκηση μας επιτρέπει να αποφύγουμε σημαντικότατες ασθένειες. Επίσης, κοινωνική πρόθεση. Μέσω του αθλητισμού μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την εκπαίδευση και την παιδεία σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και κατά αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τις κοινωνικέ ανισότητε. Έπειτα, sport business, οι επιχειρήσεις ε, του αθλητισμού, 146 δισεκατομμύρια δολάρια σε ε, παγκόσμιο επίπεδο α, εκπροσωπεί η νέα αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ασχολούμεθα όμως και με τα κακό κείμενα δραστηριότητας αυτής, όπως για παράδειγμα οι καταχρήσεις στα στημένα παιχνίδια κτλ. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να προωθήσουμε νέες νομοθετικές δραστηριότητες εμπλέκοντας οργανισμούς, επιχειρήσεις, αθλητές και διάφορους φορείς. Στις 30 Ιουνίου είχαμε την πρώτη μα συνεδρίαση παρουσία του Επιτρόπου Ναύρατζικ, ο οποίος μας παρουσίασε τις προτεραιότητές του για τα πέντε επόμενα χρόνια. Μάλλον θα λάβει χώρα τον Ιούνιο αυτή η συνεδρίαση και έπειτα το Σεπτέμβριο θα αναφερθούμε περισσότερο στον διορισμό των μεγάλων αθλητικών γεγονότων σε διάφορες πόλεις και χώρες. Η σημερινή ακρόαση σίγουρα θα επηρεάσει και τις εργασίες της δικής μας της Επιτροπής, του δικού μας του Intergroup και τα όσα θα πούμε το Σεπτέμβριο. Ήδη 4.000 άτομα από τον Νεπάλ κυρίως έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κατάρα πολύ περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές, πολύ περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό του 2022. Σίγουρα λοιπόν οι σημερινέ συζητήσει θα επηρεάσουν πάρα πολύ τι εργασίε του δικού μα, του Intergroup, το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί με όλε τι πτυχέ του αθλητισμού. Γιατί όπω σα είπα, ο αθλητισμό απασχολεί 190 εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε σε καθημερινό επίπεδο, οι οποίοι περιμένουν πολύ περισσότερα πράγματα και όχι απλώ μια επιφανειακή προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ζήτημα του αθλητισμού. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και τι δύο επιτροπέ για τη διοργάνωση αυτή τη ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Βένταρα έχει τώρα το λόγο, μέλος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και είναι μέλος, όπως το ακούσαμε μόλις τώρα, του Προεδρείου της Διακομματικής Ομάδας για τον Αθλητισμό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πρώην ε, αθλητής είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε πολλές ε, ε μεγάλες αθλητικές ε, εκδηλώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου που και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πληροφορίες που μας δώσατε, που ε, επιβεβαιώνουν τα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό. Δεν είμαι αντίθετο με αυτά που λέτε, αλλά θέλω να θέξω κάποια θέματα. Πρώτα θα πρέπει να μιλήσουμε για τον οικονομικό ε, παράγοντα. 5,7 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι η συμβολή του αθλητισμού. Ε, βεβαίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, ε, οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων, οι εμπειρίσμου μου από τους ε, ανθρώπους του αθλητισμού που από αθλητές μετά γίνονται προπονητές, Ποιο είναι ο δικό τους ρόλος σε τέτοιε μεγάλε διοργανώσει. και μια ερώτηση προ όλου σα. Ξέρουμε ότι τα έθνη θέλουν και φιλοξενούν ε, τα γεγονότα. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι η FIFA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι μόνο διεθνείς ε, ομπρέλες και ότι και οι εθνικές ε, αντίστοιχες οργανώσεις είναι πολύ σημαντικές. Οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κανόνες τους ώστε να δεσμεύσουν τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις και εθνικές επιτροπές, πράγμα που σημαίνει ότι οι κανόνες που ισχύουν στις Εθνικές Επιτροπές ε, πολλές φορές φαίνεται να είναι αντίθετη με την Εθνική Νομοθεσία. Μήπως αυτές οι εθνικές λοιπόν ε, οργανώσεις, ολυμπιακές οργανώσεις, ε, οι, οι διοργανωτές του παγκόσμιου κυπέλου, οι τοπικοί, οι εθνικοί δεν έχουν μεγάλη επιρροή. Ποιες ε, είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι που πρέπει να πληρούν τα υποψήφια κράτη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. με, εξέπληξε κάπως τα όσα είπαν τα, η εκπρόσωπος της FIFA με τα όσα είπε, γιατί αν κατάλαβα κατάλαβα καλά, ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται είναι ο δείκτης ε, ε, ε, ανάπτυξης. Και για τους υπολείπους να σας ευχαριστήσω. Και για τον κύριο Μπάουρ, για το Κατάρ και για το τι συμβαίνει με τις θέσεις εργασίας. Πολλές πληροφορίες σε σχέση με δημοσιογραφικές πηγές για να δειχθεί τι γίνεται παράλληλα με τον αθλητισμό. Όπως πολλοί είμαστε φίλοι εδώ, αλλά ανησυχούμε όπως και εσείς όταν συντάσσονται τέτοια δημοσιεύματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντζέρη, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής απέναντι στους συνομιλητές μου για να τους ε, εγκαλέσω να σκεφτούν και να μου απαντήσουν. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δυσκολεύονται στον αθλητισμό. Γιατί ε, ακριβώς οι πολιτικοί αποφάσισαν να κάτσουν στον πάγκο κάνοντας λάθος. Και αυτή η υποτιθέμενη αυτονομία και ουδετερότητα των αθλητικών οργανώσεων τελικά έχει μεταφραστεί σε αυταρχία και αυτοέλεγχο. Υπάρχει απουσία ελέγχου και οδηγιών που οδήγησε σε οικονομικές καταστροφές και σε εκτεταμένη διαφθορά καθώς και στην αποκλεισμό όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και του διεθνούς δικαίου πολλές φορές. Και όπως είδαμε και πρόσφατα, ο αθλητισμός χρησιμοποιείται όλο ένα και περισσότερο σε ένα είδος ε, ξεπλήματος συνειδήσεων, ε, μάλλον πλυντηρίου συνειδήσεων από τις κυβερνήσεις. Και το λέω στους εκπροσώπους τόσο της ΦΥΘΑ όσο και της ε, Διεθνούς Ολυμπικής Επιτροπής ως ότι η σιωπή σημαίνει συνένεση. Δεύτερο θέμα είναι ένα τεράστιο όγκο χρημάτων που μας κάνει να ξεχνάμε όχι μόνο τις θετικέ στοιχείες του αθλητισμού, αλλά και προδίδει το πνεύμα του συνεδρίου της σύσταση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής του 1984 και του χάρτη που συστάθηκε τότε και για την πολιτική. Υπάρχει ένα είδος ε, πολιτικής αποσύνδεσης της κοινή γνώμης, δηλαδή των πολιτών, των συμπολιτών μας, που εύκολα δεν κάνουν εκπτώσεις ε, στην αθλητική συνείδηση, πράγμα το οποίο δεν ε, επιτρέπουν στην υπόλοιπη δημόσια ζωή. Η πολιτική λοιπόν στην ε, νομοθετική τη διάσταση θα πρέπει να θέσει το θέμα ε, του πώς θα, όχι θα κατέβει στο γήπεδο, αλλά να ορίσει πιο συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα καταρχήν. Ε, η δεύτερη υπόθεση είναι να δώσουμε μια μεγαλύτερη ισχύ στην ε, λειτουργία της θετικής ειρήνης, ας πούμε, παιδεία, δημοσία υγεία, ε, ε, ηθική κτλ. Και τέλος, ίσως θα είναι και χρήσιμη μια εκστρατεία μεγαλύτερη ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον πολυκεντρικό χαρακτήρα του αθλητισμού και για τις συνέπειες της έλλειψης και της στήριξης των δικαιωμάτων ή του δικαίου. Ε, συμφωνώ με την κυρία Βέτ Μαΐρ σε σχέση με το θέμα του σπόρου και της εξωτερικής πολιτικής. Να θυμίσω μια, μια ε, αξέχαστη συνάντηση ανάμεσα στον Νίξον και τον Μάο Τσετούγκ το 1972 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πινκ πονγκ στην Ιαπωνία που θυμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στις, ότι στήριζε δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών η διοργάνωση αυτού του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παντζέρη και τώρα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ζαγοράκη που είναι και εκείνος σπουδαίος αθλητής. Πολύ μας ευχαριστεί να ακούσουμε έναν, τη φωνή ενός παίκτη, ενός αθλητή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, εμείς λειτουργούμε σαν ομάδα. Ε, η, η, ομάδα μας ηγείται από δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες των πραγμάτων, τον κύριο Καραμπέλα και τον κύριο Φίσας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους σας για την ενημέρωση που μας κάνατε. Πραγματικά ακούσαμε κάποια πράγματα που ε, όχι ότι ήταν περίεργα, απλά δεν περιμέναμε να έχουν, να έχουν πάρει τόσες μεγάλες διαστάσεις. Ε, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, απλά θα ήθελα με ανυπομονησία να δω την έκθεση, αυτό που είπα την έκθεση της FIFA, ε, τι έχει να πει και θα μας εκπλήξει ευχάριστα. <clears throat> Καταλαβαίνω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η θέση της, γιατί εγώ ξέρω και αυτό που από μικρό παιδί που έχουμε ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ότι οι ανθρώπινες ζωές είναι πάνω απ' όλα. Και που συμβαίνουν για να λέγονται αυτά τα πράγματα ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες νεκροί από τον Νεπάλ νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Και το ποδόσφαιρο και αθλητικός γενικότερα αυτό που μας έχει διδάξει είναι πάνω απ' όλα ήθος. Ευχαριστώ. Grazie. Eh, la collega Locke Biller, prego. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους ε, όσους παρενέβησαν. Τρεις παρατηρήσεις για την ανάληψη αθλητικών εκδηλώσεων, για το Κατάρ και πάλι και τέλος για μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτη παρατήρηση. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω στην ανάληψη τέτοιων εκδηλώσεων οι μεγάλες ενώσεις, αθλητικές ενώσεις και οργανώσεις να απαιτήσουν βελτίωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ένα θέμα ε, προς ε, τους ε, εκπροσώπους Φεστ και Τάισεν και προς την FIFA. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, πολύ συγκεκριμένες αξιολογήσεις γίνονται σε τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικού χαρακτήρα θέματα. Πώς έχει το δίκτυο των σιδηροδρόμων, ποια είναι η αξιοπιστία και τα λοιπά από ενός κράτους. Η δική μου πρόταση θα ήταν να υπήρχε βαθμολόγηση σαφής μετρήσιμων κοινωνικών και νομικών ε, παραμέτρων που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, Press Freedom Index, ε, ο δείκτης ε, της ελευθερίας του τύπου ή ε, οργανώσεων όπως της Human Rights Watch ή της Amnesty International. Να υπάρξει βαθμολόγηση τι γίνεται σε αυτές τις χώρες συγκεκριμένα με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κατά τη χρονική στιγμή πριν από την ανάληψη τέτοιων εκδηλώσεων θα μπορούσε να δοθεί ένας βαθμός, μια βαθμολόγηση και αυτός να λαμβάνεται υπόψη για την ανάληψη ή όχι από αυτές τις χώρες αυτών των εκδηλώσεων. Για παράδειγμα και για τη FIFA για παράδειγμα. Η συγκεκριμένη κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε μια χώρα είναι η πιο πραγματιστική και ρεαλιστική προσέγγιση για μια χώρα αν θέλουμε κάτι να πετύχουμε και όχι γενικόλογες προδιαγραφές για το ήθος, την ηθική που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Δύσκολο. Θα ε, Δεύτερον, θα συμφωνούσατε με μια impact assessment, μελέτη επιπτώσεων. Δηλαδή, πώς βαθμολογούνται οι επιπτώσεις σε μια τέτοια χώρα. Για παράδειγμα, για τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ ή αυτά τα οποία είχαμε στο, στον τύπο τον Απρίλιο ότι δηλαδή υπάρχουν κανόνες στο ακανονισμοί διατάξεις για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων στο Αζερβαϊτζάν. Τέτοια πράγματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να συμπεριλαμβάνονται. Τρίτον, πάει λίγο πιο πέρα αυτό, αλλά το επισημάνατε κυρία Βίτμαερ για τα το κύπελο στη Βραζιλία ότι δηλαδή θα πρέπει να ξαναεξεταστεί το πρότυπο που ακολουθείτε ότι μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση στο τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αποβαίνει προς όφελος του πληθυσμού σε, όλα τα, ε, σε όλες τις διαστρωματώσεις κοινωνικά και όχι στις υπερεθνικές μεγάλε ε, επιχειρήσεις που έχουν αυξημένη κερδοφορία και δεν έχουν καμιά σχέση με τη διαβίωση του πληθυσμού. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε αυτές τις προτάσεις. Δεύτερον, για το Κατάρ. Το Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο Απρίλιο απέστειλε μια αντιπροσωπεία στο Κατάρ να δει ε, από πρώτο χέρι πώς έχουν τα πράγματα επιτόπου. Ερώτηση προς την κυρία που εκπροσωπεί την FIFA. Ο εκπρόσωπος της FIFA που είχε έρθει εδώ ε, πέρυσι, σαν εκπρόσωπος του κυρίου Μπλάτνερ είχε πει εδώ συγκεκριμένα χειροπιαστά για το Κατάρ ότι είπε πιέζει ο χρόνος πια και ότι η FIFA πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να υπάρξει τήρηση και βελτίωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε αυτή τη χώρα στο Κατάρ. Τώρα έχουμε την έκθεση Πίπερ που κατατέθηκε και στο επίπεδο των ε, Υπουργών Εργασίας Εξωτερικών ε, στο Κατάρ που τον Απρίλιο επισημάθηκε ότι οι σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο δεν έχουν γίνει. Πολύ λίγα πράγματα υλοποιήθηκαν. Είναι δουλειά πιστεύω χειροπιαστά της FIFA η ίδια να απαιτήσει και να ασκήσει πιέσεις. Αυτά τα οποία υποσχέθηκαν να τηρηθούν και να αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στο Κατάρ. Και τα θέματα των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των εργαζομένων που δεν έχουν ε, τροποποιηθεί, δεν έχουν αλλάξει, να μπορέσουν να προαχθούν. Υπάρχουν και ε, κατηγορίες ε, για διαφθορά όσον αφορά και τη σύμπραξη από πλευράς Ρωσίας για την ανάληψη αυτής της εκδήλωσης από το Κατάρ. Όλα αυτά είναι σημαντικό να φωτιστούν. Για μας το Κοινοβούλιο τώρα τελευταίο. Ακούσαμε από διάφορες πηγές ότι πιέζει λέει ο χρόνος, ιδιαίτερα για τον Μπακού. Και υπήρξε και τοποθέτηση από μια πηγή ότι ιδιαίτερα η κατάσταση στον Πακού θα πρέπει να εξεταστεί εκ του σύνεγγης. Πρέπει να στραφούμε με, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του Κοινοβουλίου ότι το Μάιο εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλεια θα πρέπει να τοποθετηθούμε για αυτά τα κακό κείμενα στον Πακού. Αυτό θα ήταν καλό αν μπορούσε να γίνει. Και προς τις δύο συμπροέδρους μια παρατήρηση. Στο Κοινοβούλιο ποτέ δεν εγκρίναμε ένα ψήφισμα, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος, για τον αθλητισμό και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μπορούμε να μεριμνήσουμε να κάνουμε κάτι όπως η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2013, όπως τότε έγινε για το θέμα του αποκλεισμού των γυναικών. Και να πιέσουμε. Και τέλος, ε, πρέπει πραγματικά εδώ να δούμε για τις ε, π.χ. τις αθλήτριες, ε, τι γίνεται σε σχέση με τις εκδηλώσεις αυτές όταν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι από τον κύκλο των αθλητών να υπάρχουν αυστηρότερες προοπτικές για τα δικαιώματα του ανθρώπου ώστε αυτά να μην αγνοούνται πλέον. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω Για άλλη μια φορά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο και να σε ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προαναλύσαντες. Έχουμε εδώ πέρα ένα κατάλογο με διάφορα αθλητικά γεγονότα, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, στα οποία έχουν προκύψει ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή σε κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το 2012 στους αγώνες για το Αφρικανικό Κύπελο. Αλλά είχαμε επίσης και τέτοια φαινόμενα στην ε, Λευκορωσία ή ε, στους αγώνες της ε, Φόρμουλα 1. Υπήρχε στο παρελθόν δημοσιογράφος Και ως επαγγελματίας λοιπόν δημοσιογράφος σε ένα τηλεοπτικό κανάλι πριν από 10 χρόνια γνωρίζω πολύ καλά ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ορισμένες φορές αναφέρονται στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων λίγο προτού διοργανωθούν τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Αλλά βέβαια τίποτα δεν συμβαίνει, καμία δράση δεν αναλαμβάνεται αφού ολοκληρωθούν τα αθλητικά αυτά γεγονότα. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει κατά επανάληψη στο παρελθόν και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα για παράδειγμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το περσινό. Θυμάστε ότι αντί να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακούσαμε απλώς κάποιες πατριωτικές δηλώσεις υπέρ της χώρας κτλ. Οι περισσότεροι τελικά αναφέρονται στα αθλητικά επιτεύγματα, κανείς δεν θέλει να τονίσει ή να φωτίσει τη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ συχνά δεν θέλουν να πούνε τι συμβαίνει πίσω από τα στάδια, δίπλα στα στάδια, τι έχει συμβεί ουσιαστικά παρασκηνιακά. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά συνδυτή απόφαση των μέσων μαζική ενημέρωση και εκεί είναι που φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα μέσα μαζική ενημέρωση, διότι ουσιαστικά θα έπρεπε να ενημερώνουν για τα ζητήματα αυτά. Αλλά μερίδιο τη ευθύνη φέρουμε και εμεί ω Ευρωβουλευτέ. Και εμεί οφείλουμε να ενημερώνουμε του Ευρωπαίου πολίτε και εμεί πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να αλλάζουν τα πράγματα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ήδη κάποιε πρώτε πρωτοβουλίε έχουν δει το φω τη ημέρα Αναφερθήκαμε για παράδειγμα σε κάποιες πρωτοβουλίες ε, του κυρίου Λούνα Τσέκα. Ιδίω σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, της Ευρωπαϊκούς αγώνε που του Μπακού στο Αζερβαϊτζάν. Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή χρησιμοποιεί πλέον κάποιους ε, όρους, κάποιες προϋποθέσεις, τις λεγόμενες ανθρωπιστικές ρήτρε όσον αφορά την, ε, τον καθορισμό της χώρας που θα αναλάβει τους ε, επόμενους αγώνες. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να πράξει και η FIFA και κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει και με τα Asian Games, τους αγώνες της ε, Ασίας. Πρέπει να σας πω ότι απογοητεύτηκα κάπως από το λόγο τον οποίο εκφώνησε η εκπρόσωπος της FIFA θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και νομίζω ότι το είπε πραγματικά η εκπρόσωπος ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ειλικρινά με σόκαρο, οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Μας είπατε ότι πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Μας είπατε ότι πρέπει να είμαι ρεαλιστές. Μας είπατε ότι συνδιαλέγεστε με κυρίαρχα κράτη. Συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι πολύ συχνά τα κυρίαρχα κράτη μπορεί να είναι και απολυταρχικά κράτη. Ανταυτού τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά, είναι παγκόσμια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα συγκεκριμένων κυρίαρχων κρατών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καθολική ισχύ, οικουμενική ισχύ. Και αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε έθνη κράτη τα οποία χρησιμοποιούν τον αθλητισμό, χρησιμοποιούν του αγώνε, προκειμένου να καταφέρουν να αναβαθμίσουν το διεθνέ προφίλ, το διεθνές προφίλ του. Ει βάρο πολύ συχνά των ίδιων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα κίνητρα τα οποία δίνονται πολλέ φορέ. Ποια κίνητρα δίνετε εσεί όμω ω FIFA στι χώρε αυτέ. Μήπω θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα τέτοια κίνητρα για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένε χώρε. Και μα είπατε και αναφέραμε πάντα στην εκπρόσωπο τη FIFA ότι θα αναβαθμίσετε μετά το 2016 τα κριτήριά σα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι ποιο σημείο όμω μπορείτε να φτάσετε, μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε για το τι προτίθεστε να κάνετε, μπορείτε να μα δώσετε αν μη τι άλλο μια κάποια περιγραφή τη αναθεώρηση αυτή τη προσέγγιση σα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θέλω τώρα να κάνω κάποιε συγκεκριμένε παρατηρήσει. Πρώτον, εμείς ως Ευρωβουλευτές, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, πώς μπορούν από την άλλη τα κράτη-μέλη να ασκήσουν πίεση σε διεθνείς ομοσπονδίες αθλητισμού, προκειμένου οι φορείς αυτοί να θέσουν στην πρώτη γραμμή το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόσο κατά την προετοιμασία της διαδικασίας υποβολής προσφορών και διορισμού πόλων και κρατών, αλλά και κατά τη διάρκεια της δεξιαγωγής των αθλητικών γεγονότων. Όσον αφορά τώρα το μποϊκοτάρισμα, Μήπως θα έπρεπε ορισμένα κράτη να μποϊκοτάρουν αθλητικά γεγονότα τα οποία διοργανώνται σε χώρες που έχουν πολύ κακές επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μήπως θα έπρεπε να καταλήξουμε σε μια τέτοια προσέγγιση. Και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει μια τέτοια πρακτική στις εν λόγω αυτές χώρες. Και τώρα, μια πιο συγκεκριμένη παρατήρηση όσον αφορά τους αγώνες στον Πακού. Πολλοί το είπαν ήδη σήμερα, το επαναλαμβάνω κι εγώ, οι αρχές του Αζερβαϊτζάν αναμφίβολα αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα σε επικριτικούς δημοσιογράφους. Και ακόμα και αν έρθουν ορισμένοι δημοσιογράφοι και επικρίνουν όσα κάνουμε, θα τους διώξουμε από τη χώρα. Τι κάνετε εσείς για να καταπολεμήσετε τέτοιες πρακτικές. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θεωρώ και το εκτιμώ το ότι έχουμε αυτή την ειλικρινή και άμεση ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει όμως να σας πω ότι η θέση της ε, συμμαχίας των φιλελεύθερων και δημοκρατών πρέπει να μας οδηγήσει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε όσον αφορά το θέμα αυτό του αθλητισμού. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό σε αυτή την παράμετρο για μας και το, ο αθλητισμός έχει οικουμενική γλώσσα και η κοινωνία των πολιτών πράγματι στις χώρες μας παγκόσμια κιόλας κατανοεί πολύ καλύτερα τον αθλητισμό. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που πρέπει να δράσουμε άμεσα. Έχω τρεις παρατηρήσεις που θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα. Πρώτον, για τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε κάποια τεκμήρια, κάποιες μαρτυρίες κάποια χειροπιαστά στοιχεία, πληροφορίες, όταν γίνεται κάποια προπαρασκευή για την προπαρασκευή ενός αθλητικού γεγονότος σε μια χώρα και οι διεθνείς ενώσεις επιλέγουν ποιος θα αναλάβει τέτοιες εκδηλώσεις, ποια χώρα θα αναλάβει. Έχετε κάποιες πληροφορίες ότι αυτές οι αντιπροσωπείες π.χ. για τους οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητοι επαΐοντες, ε, πραγματογνώμονες, δημοσιογράφοι, που γνωρίζουν το τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες ε, και είναι και γνωστοί και υπάρχουν και αρκετά τεκμήρια, μαρτυρίες ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο ευαίσθητη και φλέγουσα εκεί. Και όταν βρίσκεται υπό εξέλιξη μια τέτοια εκδήλωση αθλητική Υπάρχει κάποια αποτελεσματική επαφή και συντονισμός μεταξύ των οργανώσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των διοργανωτών ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να υπάρχει αυτή η επαφή. Δεύτερον, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να παίζουν ανάλογα με τους κανόνες που θεσπίζονται. Ποιοι κάνουν όμως, ποιοι συντάσσουν, καταρτίζουν αυτούς τους κανόνες. Ποιοι θεσπίζουν αρχές και κανόνες για τους αθλητές και τους πολιτικούς και τους διοργανωτές που πρέπει να είναι σεβαστοί οι κανόνες αυτοί από όλους και για την Ολυμπιακή Επιτροπή και τη FIFA για παράδειγμα. Υπάρχει κάτι που να θυμάστε ως περίπτωση όπου οι δικές σας ενώσεις να είχαν κάνει μια αρνητική αξιολόγηση και να είχαν διατυπώσει συστάσεις να μην γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις στη μία ή άλλη χώρα ή έχοντας την υποψία ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και η πολιτική κατάσταση σε αυτές τις χώρες δεν βαίνουν καλώς και δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές ε, και τα όσα ε, πρέπει να τηρούνται παγκόσμια για αυτά τα ζητήματα. Έχετε κάποια τέτοια ε, ένδειξη. Και τέλος, Πρόεδρε, για να μεταφράσουμε με πρακτικό τρόπο τις ανησυχίες μας, τα μελήματά μας εδώ θα έπρεπε να ζητήσουμε από αυτούς που έχουν, είναι αρμόδιοι για τη κατάτηση της έκθεσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα θέματα τα οποία εξετάζουμε εμείς τώρα και να συζητηθούν και να αναλυθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Πρώτα απ' όλα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου και τους πραγματογνώμονες που προσήλθαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Είναι του σημασία. Θα επικεντρωθώ στους αγώνες του Μπακού. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω κάνοντας κάποιο σχόλιο στα όσα έγιναν ως, ε, διατυπώθηκαν ως αιτήματα από τους προλαρίσαντες και σε σχέση και με την, Ευρωπαϊκή, με την Ολυμπιακή Επιτροπή γιατί υπάρχει εντύπωση να ε, περάσει το, να μάθουμε το μήνυμα ποιο είναι αλλά έχω επίσης την εντύπωση ότι προσπαθείτε να αλλάξετε κάτι στις ίδιες τις οργανώσεις σας. Όμως επεξηγείτε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο και γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε τι μπορείτε να κάνετε για να προαχθούν τα δικαιώματα του ανθρώπου στις χώρες που γίνονται αυτά τα πρωταθλήματα και αυτές οι εκδηλώσεις. Αυτό θα περιμέναμε από εσάς, διότι φυσικά ακούμε εδώ τα θέματα σε σχέση με, με, την πολιτική και τον αθλητισμό. Οι ε, πολιτικές εκδηλώσεις έχουν πολιτικό χαρακτήρα επειδή υπάρχει ε, ένα πολιτική, πολιτικές επιπτώσεις ε, δημιουργούνται και όταν αναφέρθηκε ότι εσείς ε, δράτε και εργάζεστε λέτε με κυρίαρχες χώρες και δεν μπορείτε να κάνετε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα λυπούμε γι' αυτό καταλήξαμε σε ένα σημείο που φτάσαμε όπου ευτυχώς τα δικαιώματα του ανθρώπου στα δικαιώματα του ανθρώπου τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας δεν είναι κάτι που βρίσκεται στο απειρόβλητο. Η διεθνής κοινότητα μπόρεσε να φτάσει σε ένα σημείο όπου ασκούνται επικρίσεις για παραβίαση και παράβαση των ε, ε, εσκαμένων και των όσων πρέπει να ε, είναι σεβαστά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά και στις χώρες μας πρέπει να γίνεται αυτό, όχι μόνο στην Αλόδαπη, αλλά αυτό αποτελεί και τμήμα άρρηκτα αυτού που η διεθνής κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προχωρήσει και έχουν καταλήξει. Δεν δεχόμαστε πια κυρίαρχα κράτη εντός εισαγωγικών να φυλακίσουν φυλακίζουν ανθρώπους ε, να, ε, όταν ε, αυτά τα θέματα έχουν ένα, μια εμβέλεια που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Είναι κάτι ίσως το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε όμως δείχνει αυτό κάτι σε σχέση με τις χώρες αυτές όπου συμβαίνουν τέτοια γεγονότα και δεν είναι στο απειρόβλητο οι χώρες αυτές. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι θα μπορούσατε να κάνετε ώστε να επηρεάσετε τα πράγματα επιτόπου χειροπιαστά ένα πράγμα που θα ήθελα να επιτραπεί σε αθλήτριες και αθλητές ε, είναι να αυτοεκφράζονται αν επιθυμούν πολιτικά, να μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα θυμόσαστε στους αγώνες του Σότσι υπήρξαν κάποιες γυναίκες ακτιβίστριες που ήθελαν να αναζωγραφίσουν τα νύχια τους στα, χρόνια της, στα χρώματα της Ήριδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επισημαίνει τις δυσκολίε, για παράδειγμα σε σχέση με τις λεσβίες και τους ομοφιλόφιλους. Δεν θα έπρεπε οι αθλητές να μπορούν να εκφράζονται επιτόπου όταν συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί δεν προχωράτε να μπορούν να το κάνουν αυτό οι αθλητές. Εκείνοι που επιθυμούν τουλάχιστον να μπορούν να το κάνουν. Πολλοί μπορεί να μην επιθυμούν να αυτοεκφραστούν εκεί, να τοποθετηθούν. Αλλά γιατί δεν τους βοηθάτε να μπορούν να γνωρίζουν ότι μπορούν να εκφραστούν όπως επιθυμούν εκεί. Και επειδή έγινε μια παρέμβαση ζητώντας ε, να αποσαφινιστεί το θέμα του μποϊκοτάζ, <clears throat> θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και από πλευράς ακτιβισμού ε, θα θέλαμε να γίνει θα προτιμούσαμε να επιλέξουμε την χρήση, ε, την διεξαγωγή αθλημάτων και τέτοιων εκδηλώσεων ώστε να υπάρξει πίεση για να ε, ε, σημειωθούν θετικές αλλαγές και μεταβολές σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ εν συντομία. Και τώρα σε, για τους αγώνες στον Πακού και εγώ με μεγάλη ανησυχία διάβασα και έμαθα ότι ήδη η κυβέρνηση εκεί στο Αζερβαϊτζάν λέει ότι η ελευθερία του τύπου πρέπει να περιοριστεί. Και βρισκόμαστε με, σε ένα διακομματικό πλαίσιο που στις 12 Μαΐου την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνεδρίαση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις εδώ για τα δικαιώματα του ανθρώπου εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να συμμετάσχει κανείς σε αυτή την εκδήλωση θα υπάρχει και μια γυναίκα παρούσα που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα σήμερα η κόρη της Λέιλα και του Αρίφ Γιουνούς η κυρία Γιουνούς βρίσκεται εδώ σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, Μινάρα. Οι γονείς της φυλακίστηκαν τον προηγούμενο Αύγουστο και βρίσκονται στη φυλακή από τον προηγούμενο Αύγουστο. Είναι ασθενής η μητέρα της, χρειάζεται ιατρική φροντίδα και είναι φυλακισμένη λόγω του αγώνα που κάνει για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Την έχω συναντήσει τη γυναίκα αυτή, τη Λέιλα, στο, κατά το παρελθόν. Είναι δύο άνθρωποι μόνο από πολλούς που έχουν φυλακιστεί. Ο, ο Τζαφάροφ είναι ένας άλλος, ένας ακτιβιστής ε, που είχε προσπαθήσει να τραγουδήσει για τη δημοκρατία και αυτός φυλακίστηκε για 6,5 χρόνια καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και ο Ίντε Γκαβαλίεφ ένας δικηγόρος για τα δικαιώματα του ανθρώπου που βοηθά τους υπέρμακους των δικαιωμάτων του ανθρώπου καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια ε, φυλάκισης και όλα αυτά επειδή ήθελαν να ε, αναφερθούν στους πολιτικούς κρατούμενους στο Αζερμπαϊτζάν και γι' αυτό φυλακίστηκαν τώρα ζητώ από εσά εσάς, Τάισεν και πιάτσις και εσάς όλους που συμμετέχετε εδώ από την, από την Επιτροπή να καταβάλλετε προσπάθειες ε, για τους αγώνες του Μπακού τον Ιούνιο που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο να απαιτήσετε από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να απελευθερωθούν ε, οι ε, κρατούμενοι συνείδησης Τζαφάροφ, οι Γιουνούς αν το κάνετε και το πείτε αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια θετική προοπτική και θα μάθουν όλοι ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι κάτι που μπορούμε να ανεχθούμε και δεν αντισταθμίζονται σε σχέση με τα να χρησιμοποιήσετε λοιπόν παρακαλώ την παρουσία των ατόμων αυτών εδώ. Να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία. Το γεγονός ότι βρίσκονται φυλακισμένοι κάποιοι στο Αζερβαϊτζάν όχι επειδή εγκλημάτισαν, αλλά επειδή αγωνίστηκαν για την ελευθερία του εκφράζεστε, της ελευθερίας της έκφρασης. Να απελευθερωθούν αυτοί λοιπόν. Αν πετύχετε τότε πραγματικά θα είχε ανοίξει μια, ένας διάβλος για να προχωρήσουμε. Πείτε μας όμως αν, είσαστε, αν έχετε τη βούληση να το κάνετε αυτό και να προχωρήσετε. Ευχαριστώ. I think with that... Ευχαριστώ. Τσίπ, παρακαλώ. Και ολοκληρώνουμε. Θεματικά, κύριε jest με z dużymi Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Ε. Αλλά όχι για πρώτη φορά στην Επιτροπή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είμαι εξαιρετικά ευτυχής που σε, αυτό, σε αυτή την κοινή ε, εκδήλωση μαζί με την Επιτροπή Πολιτισμού εξετάζουμε αυτό το θέμα. Συχνά μιλάμε για μεμονωμένες πτυχές των αθλητικών διοργανώσεων. Μιλάμε για όρους, υπό τις συνθήκες μάλλον υπό τις οποίες εργάζονται οι εργάτες που κατασκευάζουν τα στάδια. Μιλάμε για το σκάνδαλο στο Κατάρα και αυτό ήταν ένα θέμα ακρόασης και στην προηγούμενη θητεία στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν θα επαναλάβω τα όσα είπα τότε. Ωστόσο, αυτό που επίσης ήθελα να πω είναι τι γίνεται με το όσα συμβαίνουν ε, στην σκία των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Που, πράγματα τα οποία αποφεύγουμε. Δηλαδή, επισήμως ε, ε, ασβεστώνουμε την πραγματικότητα και παρουσιάζεται μία λαμπερή πραγματικότητα και οι εθνικοί οργανισμοί αθλητισμού παριστάνουν ότι όλα πάνε καλά. Μετά όμως από τα, από τα παιχνίδια, ε, οι, όσοι επισκεφθούν τα συγκεκριμένα μέρη αποκομίζουν τελείως διαφορετικές εντυπώσεις. Είναι λεπτό το θέμα ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ισότητα σε κάποια χώρα και ότι οι ίδιοι οι ε, αθλητές δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτά που βλέπουν. Κάτι ακόμα το οποίο συζητείται στην υποεπιτροπή μας, τι γίνεται με την πορνεία παράλληλα με αθλητικές διοργανώσεις, που είναι το λίκνο των παράνομων πρακτικών, είναι το κατεξοχήν επάγγελμα το οποίο είναι θύμα εκμετάλλευσης από το οργανωμένο έγκλημα. Και κάτι ακόμα. Τι γίνεται με τις επενδύσεις. Επενδύσεις σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Θέματα τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει. Τα δικαιώματα των ιδιοκτητών γης. Εκεί που κατασκευάζονται τα στάδια. Τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες αυτών των ε, γεών. Γιατί τα στάδια όλα να βλέπουμε και ξεφυτρώνουν ε, ε, με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Όμως οι ιδιοκτήτες Πώς εξαγοράζονται, απαλωτριώνονται οι διεκδησίες τους. Υπό ποιες συνθήκες. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα αναφέρονται κάθε φορά που μιλάμε για το θέμα των μεγάλων διοργανώσεων. Ωστόσο, οι απόψει της ευρύτερη κοινωνίας δεν αλλάζουν με τα όσα εμείς αναφέρουμε στι ακροάσει μας. Να πω επίσης ότι συχνά γίνονται διαμαρτυρίες στη διάρκεια αθλητικών αγώνων. Να θυμάστε τους Αμερικανούς αθλητούς που διαμαρτυρήθηκαν κατά των ε, φιλετικών διακρίσεων στους εθνικούς ε, Ολυμπιακούς για την ε, μαύρη δύναμη. Αυτό το φαινόμενο τότε αυτό το φαινόμενο τότε ήταν πολύ ισχυρό. Σήμερα όμως αντίστοιχες εκδηλώσεις δεν γίνονται. Ήταν μια πολύ ισχυρή συμβολική χειρονομία τότε για την Black Power, την μαύρη δύναμη. Ε, και όταν έγιναν ελπικοί αγώνες στην Μόσχα, κάποιοι πήγαν Κάποιοι τον μποϊκοτάρισαν τους αγώνες τότε και αυτό ήταν μια πολιτική εκδήλωση. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν ότι οι μεγάλες αθλητικές οροδιοργανώσεις είναι τελείως ασύνδετες και άσχετες με την πολιτική. Ακόμα και αν θέλουμε να κρατήσουμε χωριστά ε, το, τον αθλητισμό και θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο απολυτικός. Και κάτι ακόμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι είναι ε, ο αθλητισμός κάτι πολύ συναισθηματικό. Και εμείς θέλουμε ε, τα συναισθήματα αυτά να είναι θετικά να υπάρχει σεβασμός για την προσπάθεια την οποία καταβάλουν οι αθλητές στην προετοιμασία των αγώνων και εσείς αναφέρατε και την εξέλιξη για την ε, ισότητα. Σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν οι αθλητικές διοργανώσεις να το ε, υλοποιήσουν αυτό. Ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κύπελο στην Πολωνία και την Ουκρανία ε, κατάφερε πολλά, αλλά δεν παρέμειναν τα, η, η επίδραση δεν συνεχίστηκε, ιδιαίτερα το στάδιο στον Τζεύσκα καταστράφηκε στη διάρκεια των συγκρούσεων στην Ουκρανία. Γειτονική χώρα, χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να δείξει ε, ότι ο αθλητισμός μπορεί να επηρεάσει εξελίξεις πολιτικού χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε το εξής. Ε. Πρέπει να, δώσω Πρέπει να δώσω τον λόγο στον Προεδρείο, αλλά δεν θα μπορέσω να δώσω τον λόγο σε όλα τα μέλη του Προεδρείου. Οι πιο σημαντικέ ερωτήσει ήταν προς την Ολυμπιακή Επιτροπή και την FIFA. Θα δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συμπρόεδρό μου φυσικά, την κυρία Κώστα. Και ε, ο χρόνος πιέζει, έχουμε ξεπεράσει τα ωριά μας. Σε γνωστοποιώ τα προβλήματα αυτά για να είσαστε αλληλέγγυοι μεταξύ σα και αλληλέγγυοι προς εμένα για να μπορέσουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε. <clears throat> Να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο τη FIFA μετά σε ένα νέο εκπρόσωπο τη ΚΟΗ γιατί αυτοί οι ίδιοι αποφάσισαν ε, ότι από πλευρά ΔΕΣΠΕΡ θα υπήρχε παρέμβαση μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά θα ακούσουμε την κυρία Κώστα. Εσεί παρακαλώ πολύ σύντομα έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη και θα προσπαθήσω κυρίως να απαντήσω στα σχόλια που έκανε ο κύριος Ντέμετς Μάκερ, η κυρία Λουνατσέκο, ε, η κυρία Μπίλερ, γιατί συνδέονται μεταξύ τους. Και βέβαια λαμβάνω υπόψη μου τα όσα υπόθηκαν από τους προναλήσαντες γενικότερα. Έχουμε προσέγγιση ανθρωπιστική, το διορθώνω αυτό άμεσα. Έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, αυτή φαίνεται και στον κώδικα δεντολογίας που έχουμε και στο καταστατικό της FIFA και στα πλαίσια της υποβολής υποψηφιωτήτων για την περίοδο 2018-2022 προσπάθησα να εξηγήσω και στην παρουσίασή μου ότι υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για την ανθρώπινη κοινωνική ανάπτυξη όπου προσπαθούμε να εγγράψουμε όλες τις δεσμεύσεις του υποψηφίου, υποψήφια χώρα ή πόλη, για το τι θέλουν δηλαδή να κάνουν όσον αφορά την κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη σε σχέση με τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου και είναι σημαντικό να αφαιρθούμε στην υποψηφιότητα του Κατάρ. Το Κατάρ είχε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία όσον αφορά το γενικότερο όραμα της χώρας για το μέλλον. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη χώρα. Νομίζω ότι οι αρμόδιες αρχές του Κατάρ είναι οι πρώτες που το αναγνωρίζουν αυτό, Άρα θα πρέπει όμως να πούμε και να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη κοινωνική ανάπτυξη από τότε που δόθηκαν, που υπόθηκε ότι η χώρα αυτή θα διοργανώσει το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο τελικά μπορούμε να προωθήσουμε θετικές κοινωνικές αλλαγές, κάνοντας τη συζήτηση αυτή, κάνοντας όλη αυτή τη διαδικασία για την ε, επιλογή της πόλης που θα αναλάβει σημαντική αθλητική διοργάνωση. Όσον αφορά το ποικοτάζ, θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα θετικά, το αντίθετο μάλλον θα συμβεί. Το ποικοτάζ αντιτίθεται στις βασικές αρχές του αθλητισμού και συνεπώς η προσέγγιση μας είναι πάντα να βελτιώνουμε την κατάσταση, να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τιμωρούμε μέσω του μποϊκοτά συγκεκριμένε χώρες. Και το μποϊκοτάζ συγκεκριμένων αθλητικών διοργανώσεων στο παρελθόν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν αποτελεσματικό, δεν επέφερε αποτελέσματα. Όσον αφορά το 2026, αυτή τη στιγμή, όπω σα είπα, γίνεται μία αναθεώρηση των κριτηρίων μα. Θα ξεκινήσει ο επόμενου μήνε τη διαδικασία υποβολή προσφορών και καθορισμού τη χώρα που θα αναλάβει του αγώνε του 2026. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί το 2017 για το ποια θα είναι η χώρα που θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρωτοσφαίρου και η διαδικασία υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει μέσα στου επόμενου μήνε, κατά τη διάρκεια πάντως του 2015. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εμείς ως FIFA θέλουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε όλες εκείνες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια των συμφωνιών που συνάπτουμε με τις χώρες που διοργανώνουν τις αθλητικές αυτές διοργανώσεις. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη. Κοιτάξτε, το ανέφερα και πριν από λίγο. Να εφιστήσουμε περισσότερο την προσοχή του κόσμου στις απαιτήσει που έχουμε εμείς από συγκεκριμένε χώρες, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο που χρησιμοποιούμε υπάρχουν συγκεκριμένε πρόνοιες, συγκεκριμένε προδιαγραφές, πάντως στο μέλλον θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να βελτιώσουμε συγκεκριμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνου σε ανθρωπιστικά κοινωνικά ζητήματα και θέλουμε επίσης να δούμε αν η χώρα είναι σε θέση να προτείνει συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς θα μπορούσε να μετριάσει κάποιες αρνητικές ε, επιπτώσεις που μπορούν να υπάρχουν στα πλαίσια της διοργάνωσης του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ιδίως όσον αφορά βέβαια τα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει ήδη στα πλαίσια της FIFA μια σημαντικότατη ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, τι έχει συμβεί από την προηγούμενη ακρόαση μέχρι σήμερα. Η κυρία Λοχμπίλερ το έθεσε αυτό. Ποια είναι τα επιτεύγματά μας μέχρι σήμερα. Τι έχει γίνει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, την ακρόαση που είχαμε στο παρελθόν είχατε εστιαστεί περισσότερο στο Κατάρ. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την τοπική επιτροπή διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, που συγκεντρώνει όλες τις κυβερνητικές αρμόδιες αρχές για τη διοργάνωση της σημαντικότητας αυτής της αθλητικής διοργάνωσης. Λαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες ενημερώσεις. Ξέρουμε ότι οι κυβερνητικές αρχές της χώρας ασχολούνται με το ζήτημα αυτό. Επίσης, η ανώτατη διοργανωτική επιτροπή της, ε, του Κατάρ, ήδη από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2014 δημοσιοποίησε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία είναι δεσμευτικά για όλους τους αναδόχους έργων που έχουν να κάνουν με τη διοργάνωση των αγώνων αυτών. Επίσης, η ανώτατη αυτή επιτροπή του Κατάρ στα τέλη του 2014, το Δεκέμβριο του 2014 συγκεκριμένα, υπέβαλε την πρώτη έκθεση συμμόρφωσης που αναφέρεται βασικά στην εμπειρία που έχουν από την εφαρμογή όλων αυτών των προδιαγραφών που θα πρέπει να διέπουν όλη τη διαδικασία διοργανωτική. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε τα στοιχεία, μας αυτά, τα στοιχεία αυτά υπόψη κάθε φορά που συζητάμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ακριβώς επειδή το Κατάρ πρόκειται να δραγανώσει το το αυτό παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, θεωρούμε ότι έχει σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο και στους τομείς αυτούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιες οι κυβερνητικές αρχές της χώρας. Είναι σαφώ να συνεχίσουμε βέβαια να αποδοκιμάζουμε του τομεί εκείνου στου οποίου πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδο, να επικρίνουμε τα κακό κείμενα, αλλά από την άλλη νομίζω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε και τι δράσει εκείνε που είχε αναλάβει η χώρα προκειμένου να κινηθεί περισσότερο στη σωστή κατεύθυνση και οι τοπικέ επιτροπέ του Κατάρ και οι συνάδελφοί μα εκεί είναι σε θέση πλέον να μα δώσουν συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν πραγματικά ότι υπάρχει σημαντική χειροπιαστή πρόοδος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σαφώς, η οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθεί πλήρως, αλλά πάντως υφίσταται και θεωρούμε ότι θα οδηγήσει στα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θέλουμε και εμείς ως FIFA να δούμε. Ελπίζω με την παρέμβασή μου αυτή να απάντησα σε κάποιες από τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες που ακούστηκαν και προφανώς είμαι στη διαθεσή σας για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε και εμείς ως διοργανωτές στα πλαίσια της FIFA, αλλά και ποιες είναι οι απαιτήσει μας και οι προσδοκίες μας από τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι υποψήφιες για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Ε, τώρα για να απαντήσετε από πλευρά Σκόη ο κύριος Φέστερ παρακαλώ. Ε. Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι από πλευρά του Γερμανικής Ολυμπιακής επιτροπή που είμαι μέλος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ολυμπιακής Επιτροπής και γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά τέτοιε ακροάσεις από τη σταδιοδρομία μου. Ευχαρίστω προσήλθαμε σε αυτήν την ακρόαση. Θέλω πρώτα να υπογραμμίσω ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι μέρος της Ολυμπιακής Χάρτας και πριν από το θεματολόγιο Ατζέντα 2020 είχαμε την Ολυμπιακή, Ολυμπιακή Ατζέντα 2020, Ολυμπιακό Θεματολόγιο 2020 σε τέτοιου είδους contracts, συμβάσεις, θα, τα δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει ρητά να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σεβαστά κατά την ανάληψη εκδηλώσεων. Πρέπει όμως να πω τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν μπορούν να μετρηθούν όπως τα εξέθεσε η κυρία Λούνα Τσεκ προηγούμενα αν για παράδειγμα με 100 μέτρα μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση 100 μέτρων και αν ανταποκρίνεται ένα Ολυμπιακό χωριό σε τεχνικές προδιαγραφές τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν μπορούν έτσι να μετρηθούν. Υπάρχουν διαφορετικές απόψει για το πώς ε, διαμορφώνονται και τι συμβαίνει με τα δικαιώματα του ανθρώπου σε μια χώρα. Και δεν είναι ποτέ στατική κατάσταση σε μια τέτοια χώρα. Να θυμηθούμε τις, ε, ε, το, Ολυμπιακό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Ουκρανία. Δόθηκαν στην Ουκρανία αυτοί οι αγώνε λόγω τη επανάσταση, τη πορτοκαλί επανάστασης σε μια άλλη συγκυρία σε σχέση με την διεξαγωγή της, ε, του, Ολυμπιακού ε, ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Κάθε χώρα και κάθε επιτροπή που υποβάλλουν έτοιμα για μια τέτοια εκδήλωση και θέλουν να την αναλάβουν θέλουν φυσικά να πετύχουν, θέλει η κάθε χώρα να πετύχει μεγαλύτερο κύρος, ε, μεγαλύτερη ας το πω έτσι απήχηση για την διεθνή της θέση. Όμως έχουμε και μία άλλη όψη του νομίσματος εδώ μια σημαντική αυξημένη προσοχή που δίνεται στην ίδια την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα αυτή. Ήμουν επικεφαλής της αποστολής ε, και για, τα, ε, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και για τους Αγώνες του Σότσι και τα είδα από πρώτο χέρι όλα αυτά και φυσικά μας απασχολούν αυτά τα θέματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου στις χώρες αυτές ε. από πρώτο χέρι όπως και πριν από το Πεκίνο και στο Πεκίνο το ίδιο το έζησα και πριν από το Σότσι και στο ίδιο το Σότσι σε επαφές με οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έτσι ήρθαμε σε επαφή και με τους εκπροσώπους δικαιωμάτων του ανθρώπου στον Πακού και είχαμε και μια συνάντηση με την, ε, τον επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής ε, και με τον Γιάννη Σκοτσάντσιτς και μου και πολλών άλλων με μια αντιπροσωπεία της Human Rights Watch και με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα συζητήσαμε και είχαμε επαφές και ο ίδιος ο πρόεδρος μας και εγώ το έκανα, ήρθα σε επαφή και συζήτησα με την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν και τέτοια θέματα φυσικά τέθηκαν και προς την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν και συζητήθηκαν. Όμως ας μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στα αθλήματα κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε, δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε κοινωνικά συστήματα, να αλλάξουμε την πολιτική μιας χώρας ή της κυβέρνησης μιας χώρας. Δεν θεωρούμε ότι τα αθλήματα είναι μέσο, εργαλείο για κάποιο σκοπό το ίδιο το άθλημα, τα ίδια τα αθλήματα είναι το κύριο μέλημά μας και αναφέρθηκε και από πλευρά Τάισεν. Τι συνεισφέρει ε, η αθλητική άμυλα, ο ανταγωνισμός για τον πολιτισμό, για την ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, τα κοινωνικά θέματα. Δεν είναι εργαλείο ο αθλητισμός για πολιτικούς σκοπούς. Όχι. Φυσικά πρέπει και μπορούν οι αθλητές και οι αθλήτες να εκφράζονται. Να εκφράζονται και να λένε ποια είναι η άποψή του, όπως το ζήτησε η κυρία Λούνατσεκ, σε σχέση για παράδειγμα με παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και επιτρέπεται να το κάνουν και αυτό. Όμω δεν θέλουμε να το κάνουν. Ναι, είπατε ότι πρέπει να έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Δεν είπατε. Ε, είναι απόλυτα αυτονόητο ότι έχουν το δικαίωμα και μπορούν να το κάνουν. Είναι ελεύθεροι πολίτε οι αθλητέ μα, οι αθλητέ που μπορούν να εκφράζονται ή και να σιωπούν αν επιλέγουν. Δεν θέλουμε όμω αυτή η πολιτική αντιπαράθεση να διεξάγεται στα γήπεδα ή στα πεδία ε, της η ομάδα για παράδειγμα του Ισραήλ όταν συναντά την ομάδα του Ιράν δεν θέλουμε η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να εκραγεί εκεί και να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην αθλητική αυτή αντιπαράθεση ή άμυλα. Καθένας πρέπει να υπομίζεται την ευθύνη του. Και αυτό πρέπει να το κάνει ο αθλητισμός και γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Ανησυχούμε κιόλας και το είπαμε αυτό και από πλευρά ε, Μίκη το γνωρίζει και έχουμε συζητήσει και συζητήσει και με πολλέ οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όμως, από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, τώρα πραγματικά δεν θέλω να περάσω το μουντζούρι σε κάποιον και να τον κατηγορήσω εκείνο να πληρώσει τα σπασμένα θα μπορούσα να πω να πάτε εκεί όπου είναι 100% διασφαλισμένα τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ε, τότε πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα σύμφωνο, για μια συμφωνία για τα ενεργειακά προϊόντα με το Αζερβαϊτζάν Αυτά τα ίδια αιτήματα διατυπώνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαπραγματεύεται με το Αζερβαϊτζάν Εδώ έχουμε και οικονομικά συμφέροντα και υπάρχουν πολύ ισχυρότερες δυνάμεις και που είναι πολύ πιο αποτελεσματικές για να επηρεάσουν επηρεάσουν κάποια πράγματα από ότι μια ένωση αθλητική ή μια οργα... Ε, διο... Ε, ένας οργανισμός αθλητικός. Ναι, ο αθλητισμός είναι πολιτικού χαρακτήρα, δεν είναι απολιτικός, το ξέρουμε αυτό. Τα, οι αγώνες διεξάγονται σε μια, σε μια συγκυρία πολιτική όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον από ό,τι στο παρελθόν. Και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αυτό και θα γίνει αυτό. Και είμαστε υπέρ του να γίνεται και να, να γίνει αυτό. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τις δράσεις αυτές. Όμως σκεφτείτε και προβληματιστείτε μια στιγμή. Ο αθλητισμός μέσα σε μια συγκυρία τι μπορεί να ε, προκαλέσει, ή να δημιουργήσει. Τουλάχιστον στην κεντρική Ευρώπη κατά το παρελθόν έγινε λόγος για το Θιβέτ τόσο έντονα και αυτά τα θέματα βρέθηκαν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και στα πιο ε, δημοφιλή ε, ε, μέσα αυτό έχει φυσικά ένα ρόλο που ε, συναρτάται και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ε, που διεξήχθησαν στο Πεκίνο τότε. Και τώρα με τους αγώνες ε, στο Αζερμπαϊτζάν τα δικαιώματα του ανθρώπου θα συζητηθούν και βρίσκονται υπό συζήτηση και εξέταση και σε κάθε εύρος και με κάθε εμβέλεια πανευρωπαϊκά. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που κάθε κυβέρνηση που ασχολείται και υποβάλλει υποψηφιότητα για αθλητικές εκδηλώσεις και η Γερμανία με το Αμβούργο θέλει να είναι υποψήφια για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Αμβούργο το 2024 πρέπει να τίθεται ο δάκτυλος επί του τύπου των ύλων και να συζητώνται αυτά ανοιχτά. Ευχαριστώ. Και για τους πολιτικούς κρατούμενους τι λέτε. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να απελευθερώσουμε πολιτικούς κρατουμένους δυστυχώς. Ξέρετε, ξέρετε, είμαστε ως ε, Ολυμπιακή Επιτροπή, είμαστε φιλοξενούμενοι στο Αζερβαϊτζάν. Και αυτή η πρώτη, ας το πω, έκδοση των European Games που θα, ε, θα διεξαχθεί εκεί και σε εσωτερικές επαφές με την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν αναφέρονται και θίγονται όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ έχω τοποθετηθεί, αλλά ας μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και την επιρροή μας είναι πολιτικούς, ε, πολιτικό ζήτημα που από τους πολιτικούς θεσμούς ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί. Για παράδειγμα από το Ευρωκοινοβούλιο, από θεσμικά όργανα, όπου δεν μπορεί κανείς να ζητά υπερβολικά πολλά πράγματα από τον αθλητισμό και τους οργανωτές του. Αν επιτρέπετε θα απαντούσατε συγκεκριμένα στην ερώτησή μου. Σας ρώτησα και είπατε τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι στατικού χαρακτήρα. Κινούνται, βρίσκονται εν ρευστό και μεταξελίσσονται. Και για το, την πρότασή μου για βαθμολόγηση, η συμπερίληψη βαθμολόγησης, ανέφερα το Press Index, όπου υπάρχει μια βαθμολογία προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν μπορείτε να αναφερθείτε συγκεκριμένα στην πρότασή μου, στην ανάληψη τέτοιων εκδηλώσεων παράλληλα με τα τεχνικά και οικονομικά οικονομικά ζητήματα, τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου να μπορούν να βαθμολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη θα έλεγα προσπαθώντας να απαντήσω και θα ζητούσα και ο αντιπρόεδρος μας να πει και εκείνος δυο λόγια διότι απάντησα σε αυτό το ερώτημα ήδη εγώ. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι μαθηματικά αριθμητικά βαθμολογήσιμο αν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, από μια χώρα ή όχι εν μέρη βρίσκονται κάποιες χώρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πώς μπορεί ο αθλητισμός και οι οργανώσεις του να αποφασίζει πόσοι βαθμοί θα δοθούν, πόσα μόρια μιας βαθμολογίας ε, θα δοθούν σε μια χώρα ή όχι και να πούμε α, δεν πρέπει να δίνονται κάποιοι αγώνες ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες επειδή εκεί ασκείται ακόμα, εκτελείται η θανατική πηγή. Αν θέλετε να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο να απαντήσει εκείνο. Παρακαλώ, ναι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. θα μιλήσω αγγλικά, θα προτιμούσα να μιλήσω την δική μου τη γλώσσα, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι της Σλοβενίας εδώ. Καταρχάς να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την πρόσκλησή σας και πραγματικά πρόκειται να διαβιβάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας στην εκτελεστική μας επιτροπή. Δεν είμαστε εμείς βέβαια μια επιτροπή που λαμβάνει αποφάσεις, είμαστε απλοί εκπρόσωποι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, Νομίζω ότι κάνουμε μια καλή δουλειά αυτή τη στιγμή. Επιτελούμε ένα θετικό έργο. Ο αθλητισμό αποτελεί τμήμα τη κοινωνία των πολιτών. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Αν για παράδειγμα φέρνουμε σε μια χώρα 6.000 ε, αθλητές, 1.300 και πάνω δημοσιογράφους, ανοίγουμε ουσιαστικά περισσότερο τις χώρες αυτές στη δημοκρατία, συμβάλλουμε στον εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών. Πάντως δεν είμαστε πολιτικοί φορείς. Δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά μας και δεν έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες όσον αφορά τον πολιτικό τομέα. Οι χώρες στις οποίες αναφερθήκατε είναι χώρες που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή είναι χώρες που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή βρίσκονται ακόμα και στο Προεδρείο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Αζερβαϊτζάν, αυξάνει όλο και περισσότερο τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες αυτές έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί τομεί όπου οι βασικές αυτές ιδέες, τα βασικά αυτά ζητήματα έχουν συζητηθεί και μπορούν να υποβληθούν συγκεκριμένε προτάσεις. Εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε πολιτικές δεσμεύσεις. Ο αθλητισμός θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και θα πρέπει ουσιαστικά να είναι και Βέβαια, εμείς θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να προωθήσουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα υποβάλουμε συγκεκριμένε εκθέσει στη δική μα Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά τη θα σε επαφή με τι αρμόδιε αρχέ του Αζερβαϊτζάν. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι λειτουργούμε. το να καταφέρουμε εμείς να υποσχεθούμε, να δεσμευθούμε ότι θα πετύχουμε συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα, πολλές φορές ακόμα και ποινική φύσης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αναλάβουμε ως υποχρέωση. Θεωρούμε πάντως ότι επιτελούμε ένα πολύ θετικό έργο, εκπροσωπείται εδώ πέρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς εκπροσωπούμε 50 κράτη της Ευρώπης, Στην πράξη, είμαστε η τελευταία όμω η οποία διοργανώνει τέτοιε ευρωπαϊκά, τέτοιες ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκούς αγώνες. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί όσον αφορά τα ζητήματα του αθλητισμού. Έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις όσον αφορά τους θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διοργάνωση από εμά αυτών των αγώνων θα συμβάλλει πάρα πολύ στον εκδημοκρατισμό, όπως σας είπα, συγκεκριμένων χωρών και νομίζω ότι είμαστε θέση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε τις ε, χώρες αυτές πιο ανοιχτές και αποτελεσματικές κοινωνίες. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο λόγια, δύο σκέψεις θα εκθέσω και μετά θα δώσω τον λόγο στην Πρόεδρο Κώστα για να κλείσει αυτή τη συνεδρίασή μας. Όχι, δεν γίνεται. Βρισκόμαστε μισή ώρα εκτός χρόνου. Λυπούμε πάρα πολύ και δεν μπορώ να δώσω τον λόγο. Λυπούμε και στην ε, Επιτροπή γιατί ε, έχουμε περάσει κατά πολύ το χρόνο μας. Εδώ κάποιες σκέψεις πολύ σύντομες. Η πρώτη, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Όχι, καθόλου. Όχι. Η πρόσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι υποχρέωση, οικουμενική παγκόσμια υποχρέωση δεν είναι μια πολιτική δραστηριότητα η δράση. Το να υπερασπίζει κανείς ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων, όλων των ατόμων, των πολιτών, των κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων, των θεσμικών φορέων, αλλά και όλων των υπολείπων. Άσχετα αν είναι διεθνείς οργανισμοί ή διεθνείς ενώσεις ποδοσφαίρου ή μια οργάνωση για κάποιο άθλημα ή κάποιου καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Είναι οικουμενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προάσπιση τους ανήκει σε όλους. Είναι οικουμενικού χαρακτήρα. Και δεύτερον, η ουδετερότητα, η αμεροληψία δεν υπάρχει. Λάθος αυτό. Διότι όχι εσεί που είσαστε εκπρόσωποι απλοί, αλλά τα εκτελεστικά όργανα. Όταν εκείνα αποφασίζουν ότι θα διεξαχθεί μια μεγάλη εμβέλεια αθλητική εκδήλωση κάπου ή ότι θα γίνει για στο Κατάρ για παράδειγμα ε, ή στον Πακού ή στο Κατάρ αποφασίζουν για κάτι που έχει τεράστια εμβέλεια αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση τεράστιας εμβέλειας και επίπτωσης και δεν θα αναλύσουμε εδώ γιατί λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις για μια τέτοια έδρα όπως το Μπακού ή το Κατάρ ή, ή άλλη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Μεταξύ αυτών των λόγων για να επιλεγεί η μία έδρα ή η άλλη που είναι μια πολιτική απόφαση πρώτου επίπεδου, ανώτατου επίπεδου, εσείς εισάγετε ως κύριο στοιχείο θα πρέπει να εισάγετε τα δικαιώματα του ανθρώπου και τίποτα άλλο παραπέρα. Και ε, σε σχέση με το δεν μπορούν να μετρηθούν, μπορούν να μετρηθούν κύριε και είναι σαφέ ότι μπορούν να μετρηθούν αν είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι και αρκετά εύκολο να μετρηθούν. Υπάρχουν συστήματα για τη μέτρησή τους. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν για την λήψη πολιτικής απόφασης να γίνουν κάποιοι αγώνες στον Πακού για παράδειγμα ή στο Κατάρ ή να διεξαχθεί το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό σε κάποια συγκεκριμένη χώρα εσείς ε, να έχετε το κύρος και την εξουσία να λαμβάνετε μια τέτοια πολιτική επιτροπή αλλά στη συνέχεια να μην επομίζεστε τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής απόφασής σας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εμείς ζητούμε βοήθεια να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων παγκόσμια που έχει, να κάνει, ε, που έχει σχέση με τη ζωή και την, ε, το σεβασμό των ανθρώπων. Και όταν οι εκπρόσωποι της Human Rights Watch, όταν κάποιος πάρει τη θέση του σε ένα στάδιο υπό τις, τα κάγκελα ε, του οποίου σταδίου αποβίωσαν δούλοι, δουλοπάροι και εργαζόμενοι, ήλωτες που ε, σκοτώθηκαν εκεί, αυτό σας αφορά και ως Επιτροπή και αφορά όλους μας και πρέπει να μας απασχολήσει. Μπορούμε να υιοθετήσουμε λοιπόν μια ψυχρή πραγματιστική θέση να πούμε «Α, δεν έχει καμιά σχέση ο αθλητισμός με την πολιτική». Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν λαμβάνετε εσείς μια απόφαση να γίνει μια αθλητική εκδήλωση στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών του χρόνου που γίνονται αυτά τα οικοδομήματα εκεί ε, υπάρχουν παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν πολιτικό ζήτημα εδώ και πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να αρθρώσουμε λόγο γι' αυτό και όχι να σιωπήσουμε. Θα πρέπει να συνεργαστείτε εσείς μέσα στις πολιτικές πρωτοβουλίες, πολλές πρωτοβουλίες που έχετε ώστε μαζί μας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις κυβερνήσεις, με όλους τους φορείς να βελτιώσουμε την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ανθρώπου παγκόσμια. Διότι είναι υποχρέωση όλων, για όλου του ανθρώπου και όχι μόνο κάποιων θεσμών. Η κυρία Κώστα, ευχαριστώ. Ε, Πάρα πολύ σημαντική η σημερινή μα ακρόαση. μα δείχνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ακόμα να εμβαθύνουμε και να τα πούμε και πιο ξεκάθαρα. Συμμερίζομαι τα όσα είπε η συνάδελφο Βαλενσιάνο, αν και καταλαβαίνω κάπω το δίλημα. Θυμίζω ότι κάποτε το δίλημα ήταν ε, αν θα συμμετείχαν ε, άνθρωποι, αθλητές ε, που έρχονταν από μη δημοκρατικές χώρες ή αν θα έπρεπε να το, στις Ολυμπιάδες ή αν θα έπρεπε να τους βοηκοτάρουμε. Γιατί τότε όμως η Διεθνής Επιτροπή ε, έλαβε αυτή την, ε, ε, προέβη μάλλον σε αυτή την επιλογή, δηλαδή να μην τιμωρήσει διπλά τους αθλητές, δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός έχει μεγάλη αξία εκδημοκρατισμού. Σήμερα όμως το δίλημα είναι διαφορετικό και καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, το έλεγε ο συνάδελφος Πανσέρη, καθορίζεται από οικονομικά συμφέροντα και το λέω ειλικρινά, το καταλαβαίνω. Συχνά έχουμε την αίσθηση ότι αυτό επικρατεί έχει γίνει βέβαια πρόοδος με τον Ολυμπιακό Χάρτη, με την Ατζέντα 2020, με τις συμβάσεις των ε, πόλων ε, υποδοχή. Υπάρχουν περιθώρια για και άλλη βελτίωση, αλλά πάντως υπάρχει ε, αυτό, αυτή, κάποια πρόοδος. Υπάρχει ε, και πρέπει να είναι στη βάση των επιλογών ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις επιλογές που είναι και πολιτικού χαρακτήρα. Δεν έχουν, έχουν αξία πολιτική. Δεν είναι απαραίτητο θεσμικά πολιτική απόφαση λοιπόν ε, αυτή η θετική συνεργασία ανάμεσα στις δύο επιτροπές μας, ε, οι οργανισμοί που ε, δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση και οι οργανισμοί οι αθλητικοί μπορούν να αποτελέσουμε ένα βήμα για να κάνουμε περισσότερα βήματα. Όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται. Άλλος ένας, άλλος ένας λόγος είναι ότι αυτά τα αθλητικά γεγονότα παίρνουν τεράστια δημοσιότητα και αυτό υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο, βοηθάει. Γιατί θα ήταν ίσως ενδιαφέρουσα μια μελέτη αντικτύπου, γιατί βοηθά αυτή η δημοσιότητα μια διαδικασία μεγαλύτερη διαφάνειας. Ωστόσο είναι επίση αληθινό ότι δεν μπορούμε να σιωπούμε απέναντι στα πράγματα. Τόσα συνέβησαν στον Φλωριάν εδώ και σε άλλου δημοσιογράφου που δουλεύουν στα στάδια, γιατί αυτό είναι κάτι καταφανές, προφανέστατο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να το αντιμετωπίσουμε πιθανότατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κάποιο κενό πολιτικής. Το έλεγε προηγουμένως ο Αντώνιο Παντζέρη και το επαναλαμβάνω, γιατί έχει δίκιο σε αυτό που ανέφερε και το έλεγε προηγουμένως και η Έλληνα στην αρχή, ότι μάλλον εμείς αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία διότι επικρατεί μια σιωπή. Σιωπή και της πολιτικής στις, ε, στις θεσμικές Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τη δική σας ε, αυτονομία την οποία σέβομαι γιατί και εγώ είμαι ε, ε, ε, πρώην αθλήτρια, ε, ε, την δέχομαι και την εκτιμώ την ουδετερότητα. Δεν σημαίνει αδιαφορία η ουδετερότητα. Σημαίνει όμως ότι ο αθλητισμός θα συνεχίσει να είναι ο χώρος όπου θα συναντιόνται αθλητές και που προέρχονται από χώρες που ίσως να είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους ή που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Έχει και πολιτιστική αξία ο αθλητισμός και δεν πρέπει να χαθεί αυτή, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί και ότι, δίνουμε, ότι έχουμε ηθική αδιαφορία για αυτά τα θέματα, κάθε άλλο. Τώρα, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, προτείνω λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί και να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση ανάμεσα στις δύο επιτροπές μας, γιατί πιστεύω πως είναι πολύ σημαντική η πτυχή της δουλειάς μας ε, και ε, αυτό θα συμμετέχουμε και στην ακρόαση για τον ΠΑΚΟΥ που θα διοργανώσει η συνάδελφος Λούνατσεκ. Ε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε μια, ένα ψήφισμα και στρέφουμε στους συναδέλφους της Επιτροπής Πολιτισμού ένα κοινό ψήφισμα για την επόμενη Ολομέλη ίσως να το προετοιμάσουμε που θα λέμε εμείς τα όσα λέμε και ε, εσείς λέτε και τα όσα πρέπει να πει η πολιτική. Επίσης είμαστε πολιτικοί. Να προσθέσουμε κάτι παραπάνω δηλαδή σε αυτά που εμείς θέλουμε από ε, τους αγώνες του Μπακού. Και εγώ αναλαμβάνω τη δέσμευση με την Επιτροπή μου το Σεπτέμβριο να αξιολογήσουμε τις νέες ε, σχέσεις που θα μπορούμε να, ε, μάλλον, να, τις νέες που θα μπορούμε να συντάξουμε, γιατί να μην σκεφτούμε μια τέτοια ε, έκθεση κοινή με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτά τα θέματα. Να μην αφήσουμε μόνο του τον κόσμο του αθλητισμού, αντίθετα να το συνοδεύσουμε. Πρόκειται για θεσμούς ε, και αξίες ε, πολύ βασικές και γι' αυτό και ο αθλητισμός είναι τόσο σπουδαίος για ολόκληρο τον κόσμο. Bueno, ε, Μάλιστα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας εδώ, αλλά όχι προτού ευχαριστήσουμε όλους σας το ότι ήρθατε, προσήλθατε εδώ, το ότι εκθέσατε τις ιδέες σας και απόψεις σας. Η δημοκρατία είναι εξάλλου η αντιπαράθεση διαφορετικών ιδεών και απόψεων. Ευχαριστώ για όλους για το έργο σας. Ευχαριστώ όλους σας. Και ευχαριστώ και καλή σας μέρα.